Okay, so now we are ready to give the floor. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Τόμ, που είναι η συγγήτρια για την πολιτική απασχόληση και κοινωνική πολιτική στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ, λέει κυρία Τόμ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω κάποια πράγματα για ποια είναι η, τι γίνεται με την έκθεση της Ευρωζώνης. 160 τροπολογίες έχουμε που υπευλήθησαν και μέχρι τώρα καταφέραμε να καταλήξουμε συμβαστικές και καλύψαμε πάνω τις μισές. Πολύ καλή τεχνική συνεδρία στην σημασία τη ε, συνεδριά των Σκιαδών που γίνει αύριο η πρώτη. Υπήρξαν πολλέ τροπολογίε που δημιούργησαν ανησυχίε επί του ίδιου θέματο και σωστά. Όλοι ανησυχούν για την απασχόληση των νέων, τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και πρόσβαση για τις πλέον ευάλωτες ε, ομάδες το ποσοστό εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα είναι πολύ χαμηλό και πολλές προσπάθειες παραπάνω πρέπει να γίνουν και συμφωνείτε κι εσείς οι περισσότεροι για τη διαφορά αμοιβή των φύλων και, για τη μέρημα των παιδιών. Υπήρξε ισορροπής τροπολογία συμπερίληψη ανθρώπων με αναπηρία στην αγορά εργασία. Υπευλήθησαν που αναφέρονται σε αυτά τα, και τα άτομα με μακροχρόνιες ασθένειες και ανίατες ασθένειες και πνευματικά προβλήματα, ψυχολογικές αναπηρίες. Είναι σημαντικό να αναφερθούν και αυτοί στην έκθεση για την ψηφιοποίηση και με τη μαρφώση της οικονομίας της αγοράς εργασίας ε, σημειώθηκε ότι νέες μορφής απασχόλησης μπορεί να δημιουργήσουν νέα προβλήματα Όπω πρόσκαιρε μορφέ εργασία, επισφαλεί μορφέ εργασία και πρέπει να καλυφθούν και αυτέ οι τροπολογίε, Αναφέρθηκε και ότι επενδύσει σε ανθρώπου και ανθρώπινο δυναμικό απαιτείται και διαβίου εκμάθηση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακή μόρφωση. Ένα σημείο που ήταν πολύ σημαντικό για όλου. ήταν η φτώχεια. Καλό ήταν να δούμε ότι πολλέ τροπολογίε υπευλήθησαν για την καταπολέμηση αυτή και αναφέρθηκαν στην ανάγκη κρίζωση τη φτώχεια και τη φτώχεια των παιδιών ιδιαίτερα ήταν καλό να δούμε ότι οι περισσότερες ομάδες συντονίζονται όσον αφορά την, Επιτροπή, την ε, πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική και με τα χαράς να συζητήσω τις συμβαστικές του σκιώδεις αύριο. Ευχαριστώ κυρία Συγήτρια. Και τώρα ε, οι σκιώδεις έχουν το λόγο για να συζητήσουμε τροπολογίες. ΕΛΚ ε, πρώτα, η κυρία Βόλς, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχάς την εισηγήτρια, τη Γιάννα Τούμ, πολύ καλή δουλειά που έκανα μέχρι τώρα και την ευχαριστούμε και συμβαστικές ε, τροπολογίες θα συζητήσουμε αύριο συνεδρίσεις σκιωδών. Πολύ καλή βάση για τις συμβαστικές και προσβλέπω σε εξέβρεση κοινών τόπων μου τους άλλους ε, σκιοδησηγητές και την εισηγήτρια τις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Πολλές υπήρξαν σημαντικές και είχαν στόχο τη συμπλήρωση εκθέσεω. Με τα χαρά είδα ότι πολλέ από τι τροπολογίε τόνισαν ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, ώστε να έχουμε ισότητα, πρόσβαση στην απασχόληση και να καλύπτονται όλε οι κοινωνικέ ομάδε. Να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε οικονομική και κοινωνική πολιτική που θα κινείται προ την ίδια κατεύθυνση και όχι αντίθετα, ούτω ώστε να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, είδα τροπολογίε με τα χαρά που καλούν για μεγαλύτερη δράση για την ισότητα των φύλων και να καλυφθεί η διαφορά αμοιβή των δύο φύλων είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία τη αγορά-εργασία. Το θεωρούν αυτό που οι συνάδελφοι επέβαλαν τροπολογίε που τονίζουν την ανάγκη των πολιτικών για την ψυχική υγεία στον αφορά την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική απασχόληση. Πρέπει σε όλου του τομεί να έχουμε αυτέ τι πολιτικέ. Είναι πολύ καλό για την ε, ευημερία όλων των Ευρωπαίων. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχική υγεία παρά το ότι υπάρχει κόστος οικονομικό και ατομικό και θα πρέπει να έχει προτεραιότητα το θέμα ψυχικής υγείας. Να τονίσω τη δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν για να εφαρμόσουν καλύτερε πολιτικέ πολιτικές στην ψυχική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια και καλό και για ειδικά μέτρα όπω και πρόθεση και πρόληψη ψυχική υγεία ε, και να εφαρμοστούν και ε, κάποιε πρώτερε δράσει, κάποιε. Ε, δράσεις που προφύλαξε αυτά τα προβλήματα. Η κυρία Μπίσοπ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους, λέει κυρία Μπίσοφ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Καλές οι προτάσεις της. Την ευχαριστούμε και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ακολουθούν σωστή κατεύθυνση. Προσβλέπουμε συνεδρίαση των σκιωδών αύριο. Ελπίζω να βρούμε καλές συμβαστικές. Θα είναι καλή αρχή. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα καλύτερα. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Η κυρία Πέτρα Χάντσεν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συγχαίρω την εισηγήτρια και τους κοιόδης. Χαίρομαι που όλα τα κόμματα θέλουν η κοινωνική διάσταση να ενταχθεί και να προωθηθεί αυτό το εξάμεινο. Ευχαριστώ όλους. Η κυρία Ζαλεύσκα από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ ειλικρινά την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Σκληρή δουλειά έγινε, μεγάλες προσπάθειες και θέλαμε να ετοιμάσουμε μια στρατηγική για αυτά τα θέματα. Είναι το τελευταίο έτος του δημοσιονομικού πλαισίου της Επιτροπής Juncker. Δύσκολο να αναλύσουμε ενδελεχέστερα την κατάσταση παρόλο που θα μας άρεσε. Γιατί πετύχαμε μόνο δύο στόχους. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έχουμε 10% αύξηση στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανεργία των νέων έχει μειωθεί επίσης κατά 10%. Αυτό μας δείχνει ότι οι προθέσεις μας είναι καλές, αλλά χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών, ούτω ώστε να πετύχουμε τους στόχους αποτελεσματικότερα. Κάθε φράση, κάθε τροπολογία συνεπώς είναι σημαντική. Και χαίρομαι που καταφέρουμε να πετύχουμε συμβαστικέ λύσει. Υπάρχουν δύο θέματα που θα ήθελα να υπογραμμίσω που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Πρώτα απ' όλα, εξατομικευμένη προσωπική ε, εκπαίδευση των ηλικιωμένων ατόμων. Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι το να μην συνεχίζεται η επαγγελματική ε, κατάρτιση ε, για κάποιους και όχι για όλους δεν πέτυχε τους στόχους. Θέλουμε επαγγελματική κατάρτιση, τεχνική κατάρτιση. Δεν μπορεί να έχει κανείς καλές προθέσεις για την επανάσταση 4 ή ε, ψηφιοποίηση της Ευρώπης αν δεν δούμε τι γίνεται με την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση. Προσβλέπω στη συνέχιση των εργασιών και πιστεύω ότι όλοι θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Η Σάντρα Περέιρα για την ΚΟΕ. Καλημέρα. Εξ αρχής, ε, ε, σε, αυτήν, σε ε, στο Κοινοβούλιο ήμασταν επικριτικοί όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης ε, τόσο εντός της ζώνης του ευρώ όσο και εκτός. Αυτές οι πολιτικές ε, στην ουσία επιβαρύνουν κάθε υποτιθέμενη προοδευτική πολιτική και γίνονται εις βάρος της εργατικής τάξης η οποία υποφέρει από την επισφάλεια ε, και από τη μείωση των μισθών. Γι' αυτό και οι δικές μας τροπολογίες διαφέρουν πάρα πολύ, ε, μάλλον αρκετά από αυτές άλλων ε, πολιτικών ομάδων, γιατί εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των όσων έχουν λιγότερα και όσων ζουν χειρότερα ε, θα γίνει μόνο με τη βελτίωση της κατάστασης του ευρώ με σύμφωνα ε, ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Η DG Ample από την Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Μαρτσέλο Ρανούτσι έχει το λόγο. Ή κάποιος άλλος από την Κομισιόν. Καλημέρα. Αντικαθιστώ τον κύριο Μαρτσέλο Ρανούτσι. Δεν έχουμε νέα σχόλια. Τα είχαμε εκφράσει την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει τότε ότι η έκθεση κατά την άποψή μας ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της απερχόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με τις ε, πολιτικές καθευθυντήριες γραμμές της ε, εκλογής σας Προέδρου κυρίας Βαντελάιαν. Η κυρία Ζωμή. Και εγώ να πω κάποια πράγματα όσον αφορά την έκθεση για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόληση στην Ευρωζώνη Προφανώ προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των ομάδων και των μελών τη Επιτροπή. 213 τροπολογίε κατετέθεσαν. Και είναι θέματα που άπτονται του πολίτου, διότι η απασχόληση προβληματίζει και του νέου που φοβούνται ότι δεν θα ενταχθούν στην αγορά εργασία και για του ηλικιωμένους που όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν κίνδυνο να βρεθούν στην ανεργία σε μια ηλικία που η κοινωνία του θεωρούν σαν ότι δεν είναι δυνατόν να απασχοληθούν, ότι πρέπει να απορριφθούν. Λοιπόν, δεν πρέπει να πέσουμε σε ιδεολογικές παγίδες που καμιά φορά εμφανίζονται σε τροπολογίες στην έκθεση. Υπάρχουν διάφορες στοιχείες που αναφέρονται στους μετανάστες. Θέλουμε μείωση των ισοτήτων και όλα αυτά δεν είναι αυτός σκοπός. Αν θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερο αντικειμενικό πλαίσιο και να μπορούμε να συνεθίσουμε διάφορε πολιτικέ ομάδε, πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίε για να επικοινωνούμε επί των πραγματικών δυσκολιών για την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Κατέθεσα μία τροπολογία, ε, την οποία υποστηρίζω ένθερμα, αφορά τους ε, γονείς στο, σπίτι, να λυθεί η, το πρόβλημά τους και τι γίνεται μάλλον, τι γίνεται με τη σύνταξή τους. Ε, λοιπόν, δεν μπορεί, ε, δεν μπορούν, αν έχουν αυτές τις ανησυχίες, να αφιερωθούν στην οικογένειά τους. Και η οικογένεια είναι η κυψέλη, εκεί που μαθαίνει κανείς να ζει στην κοινωνία ε, και να κινείται χωρίς εμπορικούς στόχους. Είναι η κυψέλη, είναι το κύτταρο όπου δημιουργείται η αλληλεγγύη ε, και υπάρχει επιμερισμός των αγαθών από αγάπη. Και δεν πρέπει να παρεμβαίνει υπερβολικά το κράτος θα πρέπει να εθετηθούν κατάλληλες τροπολογίες και οι πολίτες των κρατών μελών μας περιμένουν πραγματικές λύσεις και όχι ευσεβείς πόθους ιδεολογικούς ή μεροληπτικούς ε, που χρωματίζονται από κομματικές ε, σκέψεις. Ευχαριστώ κυρία Φράντσον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους κοιόδη για το εργό τους δύο στοιχεία να υπογραμμίσω σημασία που υπάρχει να έχουμε αποτελεσματική στρατηγική μετά το 2020 για την εκρίζωση της ένδυας και δεύτερον χρειάζεται συντονισμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα και ασφάλιση υγείας για τους εργαζομένους και καλύτερα στοιχεία όσον αφορά τους εργαζομένους. Αυτά ήθελα να υπογραμμίσω ε, όσον αφορά το σημαντικό αυτό θέμα. Ευχαριστώ. Άλλος που θέλει να μιλήσει για το θέμα. Όχι. Κυρία Συγήτρια, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, όπως είπα και στην αρχή. Ε, συμφωνούμε στις περισσότερες τροπολογίες. Βεβαίως, ε, συχνά αυτές οι εκθέσεις είναι χριστουγεννιάτικα δέντρα και κρεμάει κανείς ό,τι θέλει εκεί πάνω, αλλά είμαστε λίγο πολύ στην ίδια γραμμή και σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή απόφαση για τους κοιοδησίγητες. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 2 Οκτωβρίου. Τώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών, 10 λεπτών δηλαδή, γιατί 9,5 ώρα έχουμε την ψηφοφορία. να σας Dear colleagues, it's 9.30. Θα ψηφίσουμε τώρα τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Πρώτα θα ψηφίσουμε την συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 34 με ονομαστική ψηφοφορία ε, περιμένουμε για την κάρτα σας εντάξει όλοι Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβεστική 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή τροπολογία 48 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49 μέρος πρώτο. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Τώρα, περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων με τους διευθυντές των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που είναι αρμοδιότητος της Επιτροπής μας. Περιμένουμε λίγο να έρθουν οι προσκεκλημένοι μας. Λοιπόν, λίγα λόγια για να ξεκινήσουμε το θέμα αυτό. Όλοι ξέρουμε πως η υπηρεσία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για το έργο της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή μας συνήθω στέλνει δύο αντιπροσωπείες κάθε χρόνο στις υπηρεσίες αυτές. Η τελευταία ήταν το 2018 στο Σεντεφόπο και στην Όσα και το Νοέμβριο του 2018 στο ETF. Να κάνω μια σύντομη παρουσίαση των προσκεκλημένων μας. Ο κύριος Χουάν Μενέντες Βαλντές είναι διευθυντής ε, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθήκων Ζωής και Εργασίας. Καλώς ήρθατε. κυρία Κρίστα Σέντλατσεκ, ε, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στο χώρο εργασίας. Καλώς ήρθατε. Ο κ. Γιούργεν Ζίμπελ, διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της επαγγελματική κατάρτιση του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Καλώ ήρθατε. Και ο Τσέζαρε Ονεστίνη, διευθυντή ε, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο ε, Κατάρτισης του ETF και ε, Ζόρντι Κάρελ Διευθύντρια της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής η οποία ακόμα δεν έχει έρθει. Ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Ζωής και Εργασίας. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή μας που είμαστε πάλι στην Επιτροπή σας στην ναι, αυτή νομοθετική περίοδο. Αντιλαμβανόμαστε ότι καθώς ε, τα μέλη της Επιτροπής σας λίγο πολύ ξέρουν το αντικείμενο, καλό είναι να σας δώσω μια γενική εικόνα. Το Eurofound, ε, όπως σας είπα, είναι ακρονίμιο του Ιδρύματός μας. Μαζί με το SEDEFOP είμαστε οι δύο πεταλαιότερες αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από το 1975 Σύντομα να σας πω τι κάνουμε. Είμαστε η υπηρεσία εκείνη η οποία παρέχει γνώση για να βοηθήσει στην ανάπτυξη καλύτερων πολιτικών κοινωνικών, πολιτικών απασχόλησης και πολιτικών που σχετίζονται με την εργασία. Παρέχουμε βασικά έρευνα, συγκριτική έρευνα που θα είναι χρήσιμη στις διαβουλεύσεις σας για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής και εργασίας των πολιτών. Έχουμε μια τριμερή διοίκηση. Η διοίκησή μας αποτελείται από τα κράτη-μέλη, κατά κανόνα εκπροσώπους των Υπουργείων Εργασίας, αλλά και εργοδότες και εργαζόμενους και για πρώτη φορά θα έχουμε και έναν ανεξάρτητο ειδικό που θα διορίσει το Κοινοβούλιο που ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έρθει και θα μας δώσει μια άποψη για την εργασία μας. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Επιτροπή σας και σε προηγούμενες θητείες και Όπως είπα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ε, του προγράμματος εργασίας μας. Ε, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και έχετε και τις ε, πληροφορίες για το περσινό μας έργο στην ετήσια έκθεσή μας. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα όμως της δουλειάς ε, που κάνουμε και που σχετίζεται με το δικό σας πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, η πρόεδρος, η κυρία Φάντερ Λάιν, αναφέρθηκε ε, σε μια οικονομία η οποία θα αποδίδει για τους ανθρώπους η κοινωνική πτυχή της ανάπτυξης. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της ποιότητας εργασίας, δηλαδή όχι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η ποιότητα της εργασίας που είναι σημαντική. Εκεί πέρα βλέπετε λοιπόν τα σχετικά δεδομένα. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη έννοια, ένα κομμάτι αυτής είναι η μισθή. Η κυρία Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρόταση ενός νομικού μέσου έτσι ώστε να υπάρχει για τον κάθε εργαζόμενο ένας βασικός μισθός ώστε να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς ε, εκεί όπου εργάζεται και εδώ πέρα ε, στον τομέα αυτών έχουμε παράξει αρκετή έρευνα τα τελευταία έτη επίσης έχουμε εξετάσει τις ε, συλλογικές συμβάσεις εξετάσαμε πέρσι την έννοια ενός ε, αξιοπρεπούς ε, μισθού και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον τομέα. Στις 3 ε, Σεπτεμβρίου η Επιτροπή σας υπερψήφισε ενός υπέρ ενός πιλωτικού έργου για τον βασικό μισθό και βεβαίως είμαστε στην διάθεσή σας για να σας στηρίξουμε αν η Κομισιόν αποφασίσει αν εγκριθεί κάτι τέτοιο να ανατεθεί σε εμάς. Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά την ισότητα των φύλων όπου η κυρία Φαντελαέν ανακοίνωσε την σχετική στρατηγική και δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια ε, των αμοιβών. Έχουμε εκδώσει μία έκθεση τα τελευταία χρόνια για τις συστάσεις για την μισθολογική διαφάνεια και σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό και να κάνουμε κάποια περαιτέρω εργασία για να βοηθήσουμε την πρωτοβουλία αυτή και να βοηθήσουμε και τα νομοθετικά όργανα. Αυτό έρχεται βεβαίως μετά από πολλή έρευνα σε ζητήματα φύλου. Είχαμε πολλές εκθέσεις στον τομέα της ισορροπίας ζωής και εργασίας και στηρίξαμε κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες στην τελευταία νομοθετική περίοδο υπό τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και της σχετικής πρότασης οδηγίας για ισορροπία εργασίας και ζωής. Υπολογίσαμε το κόστος της χαμηλότερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ε, στην τελευταία ενημέρωση που κάναμε γύρω στα 30-40 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη του ότι δεν ε, υπάρχει ε, ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών που εργάζονται. Βρήκαμε μια παρόμοια μεθοδολογία που είχαμε και στο παρελθόν για τους νέους οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν εκπαιδεύονται. Ένα τρίτο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την μετάβαση, την δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και το ευρωπαϊκό ε, Green Deal και αυτούς οι οποίοι επηρεάζονται από αυτό. Μας ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πιλωτικό έργο το οποίο αφορούσε το μέλλον της βιομηχανίας και κάναμε μια πρόβλεψη ε, έχοντας και ένα μοντέλο που ανέπτυξε το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, για τις συνέπειες για μια πρόβλεψη μέχρι το 2030 ε, της εφαρμογής των μέτρων ε, της Συμφωνίας των Παρισίων και το αποτέλεσμα ε, είναι θετικό συν 1,1% αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη συν άλλο 0,5% δημιουργία θέσεων εργασίας βεβαίω αυτό είναι ένα καθαρό νούμερο δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι εκπροσωπεί πολλές αναδιαρθράσεις αναδιαρθρώσεις, με συγχωρείτε, κλάδοι θα εξαφανιστούν ε, και άλλοι θα αναπτυχθούν. Είναι ένας τομέας που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε διάφορα μέσα, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης, μια σειρά δηλαδή βάσεων δεδομένων ε, και στηρίζουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, ε, το οποίο θα συζητήσετε αργότερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο είναι επίσης ε, ένα παρατηρητήριο το οποίο παρέχει πληροφορίες για τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές ε, και για την μετάβαση από τον άνθρακα αλλά και άλλες παγκόσμιες τάσεις, την παγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση κτλ. Αυτό είναι άλλος ένας τομέας όπου έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά για τις νέες μορφές απασχόλησης επίσης, εξετάζοντας τις ε, διαφορετικές ε, συνέπειες ε, και επιπτώσεις των νέων μορφών εργασίας, οι πλατφόρμες και οι εργαζόμενοι σε αυτές, κατά το οποίο ανακοίνωσε και η Νέα Κομισιόν ότι σκοπεύει να βελτιώσει όσον αφορά δηλαδή τις συνθήκες εργασίας. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα. Όπως σας είπα, δεν θέλω να αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες του προγραμματός μας. Θα λάβετε κάποιες πληροφορίες και ένα φυλαδιάκι για το τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για εσά το πώς συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο, πώς το είχαμε κάνει στο παρελθόν. Από τις συνήθεις ακροάσεις, όπως αυτή εδώ στην Επιτροπή σας, ε, όπου ασχολούμαστε περισσότερο με την ουσία, αλλά μας έχετε ζητήσει να συντάξουμε κάποια επιπλέον έγγραφα που θα σας βοηθήσουν. Επίσης θα βρείτε τους συναδέλφους μας από το γραφείο Βρυξελών, η συνάδελφος είναι εκεί. Μια φορά θα είναι στην επιτροπή σας, θα την δείτε, οπότε χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν. Ευχαρίστω να σας διευκολύνουμε και είμαστε υπόλογοι στο κοινοβούλιο αυτό, στο διοικητικό μας συμβούλιο, αλλά πρέπει βεβαίως ε, να ερχόμαστε εδώ για να λάβουμε και την απαλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε και κάποιους δείκτες απόδοσης για να ε, σας δείξουμε ότι έχουμε αποτελέσματα σε αυτά τα οποία κάνουμε. Κάποιοι τέτοιοι δείκτες είναι το πόσες φορές χρησιμοποιούνται τα ευρήματά μας. Πέρσι ήταν σε 200 έγγραφα, 82% αξιολογήθηκαν ως έγγραφα κλειδιά γιατί ξεκινούσαν νέες πολιτικές διαδικασίες και αυτό περιλαμβάνει και κάποια ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αυτό το οποίο αφορά την ισότητα των φύλων ή το Ευρωπαϊκό Εξήμινο, εξάμεινο, η ετήσια έκθεση ανάπτυξης κτλ. Έχουμε επίσης ε, συνεισφέρει και σε διάφορες εκδηλώσεις ε, και στο Κοινοβούλιο όπου ε, έρχονται εδώ πέρα οι ειδικοί που σας δίνουν ακριβώς τα στοιχεία τα οποία χρειάζεστε. Είναι εύκολο λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί μας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας στηρίξουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για το ότι τηρήσατε έναν χρόνο τον οποίο δεν σας προανακοίνωσα, αλλά ε, νομίζω πως ε, ε, κάθε διευθυντής υπηρεσία, οργανισμού μάλλον, θα έχει 10 λεπτά για την εισήγησή του και μετά θα δώσω το λόγο σε εσά σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Σύμφωνοι. Ωραία. Και τώρα η κυρία Κρίστα Σέντλατσεκ, παρακαλώ να ακούσουμε και τη δική σας ε, εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ και που βλέπω νέα πρόσωπα και νέους ε, ε, συναδέλφου. Ελπίζω πως θα έχουμε πολύ κανή καλή συνεργασία τα επόμενα χρόνια. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας διαρκώ και πολύ θα γνωρίζετε πως Έχουμε και ένα γραφείο στις Βρυξέλλες με Οπότε μπορείτε να έρθετε πιο εύκολα σε επαφή μαζί μας. Ήθελα να ξεκινήσω με μια παρουσίαση του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είμαστε ένα μικρό μιας οργανισμός. σημαίνει αυτό ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε εκπρόσωπους ε, από τις ε, κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους όλων των χωρών. Έχουμε και μια μικρότερη ομάδα που προσπαθούμε να ετοιμάσουμε αποφάσεις και για πρώτη φορά Σύμφωνα με τον ιδιωτικό μας κανονισμό έχουμε έναν συνάδελφο, έναν εμπειρογνώμονα από εσάς που παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα θέλαμε ίσως να έχουμε και πιο συγκεκριμένες συμβολές από τη δική σας πλευρά. Είμαστε 67 άνθρωποι, στο Μπιλμπάο είναι η έδρα μας, στην Βόρεια Ισπανία και χειριζόμαστε αρκετά χρήματα. Έχουμε πάνω από προπολογισμό 15 ε, εκατομμύρια ευρώ και σε σχέση με το προσωπικό μας είναι αρκετά μεγάλο ποσό, αλλά πιστεύω πως κάνουμε καλή δουλειά. Θα δείτε εδώ στη διαφάνεια ότι είμαστε ε, μία, ε, ένας οργανισμός δικτύου, δηλαδή συντονίζουμε και ένα δίκτυο 28 εθνικών δικτύων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο απασχόλησης. Αυτό σημαίνει πως έχουμε σε κάθε χώρα μια επαφή που εργάζεται για το δικό μας οργανισμό και συντονίζει την ε, εργασία μας ε, ώστε να εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι μοναδικό γιατί αυτό σημαίνει εύκολη πρόσβαση στο εθνικό επίπεδο και εύκολη επαφή και ανταπόκριση από το εθνικό επίπεδο ε, και βέβαια συμβάλλουμε όλοι μαζί στο να διαδοθεί το σημαντικό μήνυμα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Έχουμε επίσης και ένα δίκτυο εταιριών που συνδέεται με την εκστρατεία μας για υγιή χώρο εργασίας. Είναι τεράστια αυτή η εκστρατεία. Είμαστε σε άμεση επαφή με εταιρείε για να έχουμε και τη δική του συμβολή, γιατί είναι οι πρεσβευτές μας για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αλλά και φυσικά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων συνεργαζόμαστε για να έχουμε στενή επαφή. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζετε ότι, είναι το, ότι έχουμε δίκτυο και θα δείτε και στο ε, ε site, ε, το διαδικτυακό site ποιοι είναι οι συνεργάτες μας, κυρίως είναι επιθεωρητές εργασίας, από τις επιθεωρήσεις εργασίας. Να σας πω τώρα ποιες προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί δεν, και λέω εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί δεν αφορά μόνο, αφορούν μόνο οι προκλήσεις αυτές την υγεία και την ασφάλεια αλλά και την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα ε, υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί είμαστε σε εθνικό επίπεδο, αλλά ε, θέλαμε να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, ώστε δηλαδή να πάρει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ιεράρχηση των ε, θεμάτων. Επίσης έχουμε Το γεγονός της γύρανσης ε, του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τι σημαίνει αυτό για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Πρέπει να βελτιώσουμε τα στάνταρ και τις συνθήκες εργασίας, γιατί διαφορετικά οι γυριότεροι άνθρωποι δεν θα μπορούν να εργάζονται μέχρι τα 67 ε, και στις βορειότερες χώρες μέχρι τα 70 ε, να Αναφέρω επίσης και τις μικρο, μικρές και πολύ μικρές εταιρείες που επίσης έχουμε ε, ιδιαίτερη πίεση στις εταιρείες αυτές. Ε, τώρα, ψηφιοποίηση, μια από τις προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια, στην οποία θα επανέλθω αργότερα, είναι ε, η ψηφιακή εποχή, γιατί έχουμε ειδική τεχνολογία όπου προσπαθούμε να εντοπίσουμε πιθανά σενάρια και πιθανές, ε, πιθανά προβλήματα ε, και εργασιακές ασθένειες που σχετίζονται με την ψηφιακή εποχή. Τώρα, εδώ θέλω να σας δείξω γιατί είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Βλέπουμε πως έχουμε ετησίως 150.000 θανάτους που σχετίζονται με την επασχόληση και δεν προέρχονται από ατυχήματα γιατί και έχουμε βελτιώσει την κατάσταση, αλλά σχετίζονται με ασθένειες και το κόστος είναι τεράστιο. Το κόστος αυτών των ε, νόσων είναι για την Ευρώπη 764 δις ευρώ ετησίως, 3,3 του ΑΕΠ. Δηλαδή ε, είναι κάτι όμως που πιστεύω ότι μπορεί να αποφευχθεί και να προληφθεί με τη σωστή διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Θέλω να σας το αναφέρω και αυτό εδώ γιατί είναι μια από τις προτεραιότητες. Αν δούμε τους θανάτους που αποδίδονται στην, εργασία, στην απασχόληση, οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στον δολοφόνο καρκίνο. Όχι μόνο καρκινογόνες ουσίες, αλλά και ακτίνες χ, Είναι μεγάλο πρόβλημα για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Να σας πω τώρα τι κάνουμε. Εδώ έχουμε τις προκλήσεις. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι έχουμε συμφωνήσει μαζί με τη διαχείριση την Κομισιόν και εσά το Κοινοβούλιο και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς έχουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα που είναι πολιετές και έχει παραταθεί μέχρι το 2023 αυτό το πρόγραμμα στη τελευταία μας ε, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα σας αναφέρω κάποιες από τις πτυχές του προγράμματος. Υποστηρίζουμε τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικών επί τη βάση στοιχείων. Τι κάνουμε, παρακολουθούμε μακροχρόνια και μεσοπρόθεσμα τις διάφορες δραστηριότητες. Ας πούμε υπάρχει μια έρευνα για τις ε, ε, εταιρείε για τους νέους αναδυόμενους κινδύνους. Η έρευνα αυτή λέγεται SNR, περιλαμβάνονται 33 χώρες και εταιρείε κάθε μεγέθους, ακόμα και πολύ μικρές, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση της, της παιδείας για τη βελτίωση της ασφάλειας της εταιρείας. Έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα που συλλέγουμε εθνικά στοιχεία και παρουσιάζουμε έτσι ποια είναι η κατάσταση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε ε, τους, μια, νέα, μια νέα έρευνα που ερευνά τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τον καρκίνο. Θέλουμε να συλλέξουμε εδώ όχι μόνο πληροφορίες για τις καρκινογόνες ουσίες, αλλά και για παράδειγμα συνδυασμούς ε, ουσιών σε επίπεδο επιχειρήσεων. Εργαζόμαστε επίσης για το κόστος των ατυχημάτων ε, και των ε, ασθενειών Μελετάμε επίσης ε, τις ε, μυοσκελετικές ε, τα μειοσκελετικά προβλήματα, του ψυχικούς κινδύνους, τη στήριξη για τη συμμόρφωση, δηλαδή πώς θα βελτιωθεί η εφαρμογή των στάνταρ υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και πώς θα εφαρμοστεί στις πολύ μικρές εταιρείες. Αυτό Αυτά λοιπόν σχετίζονται με τις εταιρείε. Η άλλη πτυχή είναι να στηρίξουμε τις εταιρείε με πρακτικό τρόπο, τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε δύο βασικές δραστηριότητες. Τη μεγαλύτερη εκστρατεία για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, που διαρκεί 2-3 χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ και δύο χρόνια έχει γίνει για τις επικίνδυνες ουσίες. Η επόμενη είναι οι καρδιακές παθήσεις και η τρίτη αφορά την ψηφιοποίηση και συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. σε Έχει μεταφραστεί το υλικό σε όλες τις γλώσσες. Και κάτι άλλο, ε, πολύ πρακτικό ε, θέμα για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες έχουμε φτιάξει ένα επιγραμμικό εργαλείο για την αξιολόγηση του κινδύνου. Είναι προσβάσιμο δωρεάν και υπάρχει ένας κατάλογος ώστε κανείς να μπορέσει να κάνει μόνος του αξιολόγηση κινδύνου και μετά βέβαια να δει και ποια μέτρα ε, θα πρέπει να λάβει. Αυτά λοιπόν για να δείτε τι κάνουμε και όπως είπα παρακαλώ επισκεφθείτε το, το, το website μας, είναι σε όλες τις γλώσσες, έχουμε πολύ υλικό και έχουμε και την Brenda Brian όπως σας είπα στο γραφείο επαφής μας στις Βρυξέλλες και είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ο κ. Σίμπελ, ε, ο επικεφαλής του Σεντεφόπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαι εδώ, σε αυτό το υπέροχο κτίριο. Βήκα στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ μόλις την 1η Σεπτεμβρίου. Δείξτε υπομονή απέναντί μου. Είναι η πρώτη μου παρουσίαση. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, όπως ανέφερα και οι συνάδελφοι, είναι ένας από τους παλαιότερου οργανισμούς. Ξεκινήσαμε το 1975. Προωθούμε την κατανόηση των συστημάτων κατάρτιση και εκπαίδευση, Παρέχουμε υποστήριξη και διαμορφώνουμε τη διαδικασία της Κοπενχάγης από το 2000 Πάμε σε αυτά τα θέματα μέσω της, ε, του προγράμματος για την εκπαίδευση και την παιδεία μέχρι το 2020, επαγγελματική κατάρτιση, έχουμε υποστηρίξει την υλοποίηση της σχετικής πολιτικής και παρακολουθούμε την πρόοδο που επιτελείται από το 2007. Έχουμε ε, και πιο μεγάλο ρόλο που παίζουμε για την υποστήριξη της πολιτικής και τέλος φέτος με τον αναθερημένο μας κανονισμό που ισχύει Επίσημα, έχουμε συμπεριλάβει και αναγνωρίσει δραστηριότητε που ξεπερνούν την εκπαίδευση και κατάρτιση και που εφαρμοζόταν επί καιρό, δηλαδή ανάλυση αγοράς εργασίας και δεξιοτήτων και ανάλυση προσόντων. Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ επίσης αυτά που σας είπα μόλις τώρα στη διαφάνεια και για το νέο κανονισμό μας, εσωτερικό κανονισμό, τον ιδιωτικό μας κανονισμό, αναφέρονται οι διάφοροι στόχοι μας. Όπως ανέφερα, είμαστε ένα μόνο κέντρο έρευνας ποσοτικής και ποιοτικής για την επαγγελματική κατάσταση εκπαίδευση και για τους νέους και για τους ενήλικες, δεξιότητες και προσόντα η ανάλυση μας των σχέσεων δεξιοτήτων, προσόντων και θέσεων εργασίας τώρα και στο μέλλον ε, δίνουμε πληροφορίες σε αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική για να διαμορφώνουν τις κατάστασεις πολιτικές και βοηθήσαμε στον ΤΕΦΟΠ να έχουμε πετύχει εργαλεία διαφάνειας βάσει των αποτελεσμάτων της εκμάθησης έχουμε υποστηρίξει μεταρρύθμιση στον τομέα της παιδείας και κατάρτισης μέσω εργαλείων που έχουμε δημιουργήσει και έχουμε αλλάξει και κάπως την αντίληψη που υπάρχει για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Αυτό έχει ενισχύσει και το ρόλο του οργανισμού μας. Είμαστε σημείο διαπαφή μεταξύ εκπαίδευση κατάρτιση από τη μια και αγοράς εργασίας από την άλλη. Είναι ένας τομέας που δεν καλύπτεται από άλλους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω τις προτεραιότητες του έργου μας, τη μελλοντική μας πορεία το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει πολιτή προγράμματα. Καθορίζονται αυτά από το όραμά μας που βλέπετε, από τις αξίες μας, τους πολιετής στόχους που καθορίζονται για μας και υλοποιούμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσω των τριών μας αξώνων βασικά που ακολουθούμε. Σας παρουσιάσω. Η διαμόρφωση λοιπόν του τομέα παρακολουθούμε την πρόοδο που ήταν χάνεται Ποιε είναι οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και κατάρτιση βάσει των συμπερασμάτων τη Ρήγα. Έχουμε το ReferNet, αφορά την κατανόηση των τεκτενομένων σε εθνικό επίπεδο και είναι και δίκτυο για ανταλλαγή στοιχείων και εμπειριών όσον αφορά τον τομέα. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το παρελθόν και βάσει του παρελθόντος να ενημερωθούμε για το τι θα κάνουμε στο μέλλον και ενοτομούμε όσον αφορά την παρουσίαση των στοιχείων μας από εκθέσεις που δημοσιεύαμε Τώρα πάμε σε διαδραστικά εργαλεία στο διαδίκτυο. Χαρτογραφούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί που θέλουν να μάθουν. Έχουμε ένα σύστημα βαθμολόγηση κινητικότητα, βασικέ δεξιότητε. Ξεπερνάμε την εποπτεία, διεξάγουμε, οργανώνουμε εργαστήρια με εκείνου που διαμορφώνουν την πολιτική και για αυτού ψηφιακή εκμάθηση και πολιετή δεξιότητε. Το κάναμε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Και τέλο, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ παρέχει και τροφοδοτεί εργαλεία όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, των προσόντων και το σύστημα για, τη, για, τα διάφορα, για τις γνώσεις και τις δεξιότητες και δημιουργούμε εργαλεία. Μετά, άλλος άξονας, στρατηγικός τομέας, είναι η αξιολόγηση αυτού του τομέα. Τι κάνουμε. Το ΣΕΝΤΕΦΟ προωθεί την πρόσβαση, την ελκυστικότητα και την κάλυψη επαγγελματικής κατάρτισης και παιδείας και της εκμάθησης από πλευράς ενηλίκων χρησιμοποιούμε προσανατολισμούς και αξιολόγηση και χρησιμοποιούμε κίνητρα και χρηματικά και μη χρηματικά εστιαζόμεθα επί ομάδων που χρειάζονται συγκεκριμένη προσέγγιση στα μέτρα τους για να εντάξουμε ή πανεντάξουμε στην αγορά εργασίας ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους με λίγα προσόντα και εκείνους που έχουν αποχωρήσει από το σύστημα το εκπαιδευτικό νωρί, πρώιμα. Όσον αφορά την εκμάθηση και τη μαθητεία, Διευκολύνουμε την εκμάθηση σε διάφορες χώρες και την ανταλλαγή ε, εμπειριών. Εξετάζουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των ε, δασκάλων και, και των εκπαιδευτών και το ΣΕΝΤΕΦΟ προσπαθεί να κατανοήσει τις απόψεις των πολιτών για την εκμαντική κατάρτιση και εκπαίδευση και τη διαβίωση εκμάθηση μέσω των ε, διαφόρων σφιγμομετρήσεων. Βασική ομάδα που αποφασίζει κατά πόσο ο τομέας αυτός γίνεται αποδεκτός και θεωρείται αποδεκτό για την εκπαίδευση είναι οι γονεί. Οι γονεί που αποφασίζουν για τα παιδιά του, για την επαγγελματική του κατάρτιση και εκπαίδευση. Πρέπει να πλησιάσουμε και του γονεί. Τώρα να ενημερώνουμε για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση είναι η τελευταία μα προτεραιότητα. Εδώ το ΣΕΝΤΕΦΟ παρέχει ε, ε, πληροφορίε στην αγορά εργασία και στοιχεία για να υποστηρίξει τη μετάβαση στο νέο χώρο εργασία, στο νέο κόσμο τη εργασία. Έχουμε προβλέψει προσφορά και ζήτηση για την εκπαίδευση κατάρτιση είναι μεθοδολογία που έχει δοκιμαστεί. Βλέπουμε για συνειτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο 100 μελών. αναλύουμε επίσης προσφορά και ζήτηση, τι ανισορροπίες υπάρχουν εκεί και αν δεν υπάρχει σωστή προσαρμογή δεξιοτήτων με τι ανάγκε. και επίση στο διαδίκτυο με στοιχεία τεχνολογίε big data παρουσιάζουμε τι ε, ανάγκε, τι ζητούν οι εργοδότε για να έχουμε πιο βραχή χρόνο αντίδραση αντί να έχουμε μαρκοσκελείς έρευνε που είναι παχθεί. προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και τα βγάζουμε στο διαδίκτυο να χρησιμοποιούμε λοιπόν τα στοιχεία του διαδικτύου Όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτήτων, έχουμε κάνει εκθέσει επί τεσσάρων χωρών το 2017. Είναι στην τελευταία φάση αυτέ οι έρευνε, και η διάσκεψη θα ακολουθήσει σχετική το 2020. Τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, η έρευνα για τις ευρωπαϊκές εταιρείε είναι κάτι που με κάνει υπερήφανο. Μαζί με το Eurofound ε, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και διεξάγουμε και ένα δεύτερο γύρο ε, έρευνας για τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και τις γνώσεις. Η πρώτη είναι το 2014 και συλλέγουμε στοιχεία για να λύσουμε δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης από πλευράς εργοδότη και πλευράς εργαζομένου. Εξετάζουμε το θέμα. Τέλος, με αυτές, αυτούς τους στρατηγικούς άξονες, στους που παρουσίασε, ε, θέλουμε να παρουσιάσουμε για τα αποτελέσματα, να τα προβάλλουμε, να δείχνουμε τι γίνεται, αποτελέσματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, σας δείχνω τι κάνουμε, δημοσιεύουμε πληροφορίες, ε, έντυπα, φυλάδια για τις αστηριότητές μας, όποιες ενδιαφέρεται από εσά. Έφερα και αυτό το, έχω και αυτή την παρουσίαση επίσης να σας δώσω. Ε, μετά μπορείτε να πάρετε τα έγγραφα από μένα, τα έντυπα. Το 2019 κινηθήκαμε σε αυτό το χώρο. Ε, την ανάλυση κενών θέσεων αναγκών για απασχόληση στο διαδίκτυο. Ξεκίνησε το 2018, προβλέψει αδεξιότητες, δίκτυ, τι γίνεται με τη μαθητεία, ε, βολιδοσκοπήσεις, διάφορους πόρους για να χαράσουν ανατολισμούς και αργότερα φέτος θα δώσουμε και στοιχεία για τα διάφορα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης επενδύσεων στη διάφορα κράτη-μέλη και στην ε, Νορβηγία και την Ισλανδία μέσω ενός εργαλείου που θα διατίθεται στο διαδίκτυο. Τέλος, η προτελευταία διαφάνεια. Κάποια στοιχεία για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Δεν θα φερθώ σε λεπτομέρειες. Βλέπετε εδώ στις διαφάνειες τα νούμερα για να έχετε μια ιδέα όσον αφορά τις δραστηριότητε μας και θα φτάσω στη τελευταία διαφάνεια να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις μας για το μέλλον θα αλλάξει η φύση της επαγγελματική κατάρτισης και παιδείας στην Ευρώπη θέλουμε να διευκολύνουμε την εκμάθηση να μάθουμε το παρελθόν να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες των διαφόρων επιλογών για το μέλλον τι προσπαθούμε να κάνουμε να επισημάνουμε τάσεις δεν θέλουμε να προβλέψουμε το μέλλον, τουλάχιστον όμως εκείνοι που διαμορφώνουν την πολιτική να μπορούν να ε, λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Έχουμε τρία σενάρια που αναλύουμε και ερευνούμε. Πρώτα απ' όλα πλουραλιστική προσέγγιση για επαγγελματική κατάρτιση και παιδεία. Ε, είναι το συνηθισμένο μονοπάτι για όλους. Στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης εκπαίδευσης θα εντάσσονται και στην ανώτερη παιδεία. Μετά έχουμε άλλο στενάριο που είναι συνηθισμένο, κανονικό, αλλά διακεκριμένος τομέας, διακριτός τομέας και τρίτο ενδεχόμενο σενάριο, εξειδικεσμένη εκπαίδευση και παιδεία, επαγγελματική, με στόχο τη διευκόλυνση ε, της ένταξης στην αγορά εργασίας για ειδικές ανάγκες αυτό που έχουν ειδικέ ανάγκε. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και περιμένω να ακούσω ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κ. Τσέζερε Ονεστίνη, επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την κατάρτιση του ETF, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και πάλι στην Επιτροπή σας και που μπορώ μαζί σας να μοιραστώ μια ενημέρωση για την πρόοδο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης. Θα πω δύο λόγια για όσους δεν γνωρίζετε την εντολή μας και θα περάσω γρήγορα στις δραστηριότητές μας. Το ETF είναι ένας οργανισμός ε, που έχει την εντολή να συνεργάζεται για χώρες, με χώρες εκτός της Ένωσης. Στηρίζουμε την παιδεία και την κατάρτιση και τη μεταρρύθμιση αυτών στις χώρες. Στηρίζουμε την ανάπτυξη ε, δεξιοτήτων σε χώρες εκτός της Ένωσης. Ε, ο οργανισμός μας εστιάζεται στις περιοχές της γειτονίας και της διεύρυνσης. Βλέπετε εδώ στο χάρτη ε, χρωματιστά τις κύριες χώρες συνεργασίας ε, ο βαθμό στον οποίο συνεργαζόμαστε με τις χώρες αυτές εξαρτάται στις σχέσεις που έχουν οι χώρες αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν διαφορές ε, είδη συνεργασίας και με όλες τις χώρες εστιάζουμε στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος κατάρτισης. Βλέπουμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της κάθε χώρας Έχουμε χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέση Ανατολής, την Άπο Ανατολή, Κεντρική ε, Ασία. Ε, αλλά βλέπουμε, εκεί χρειάζονται διαφορετικοί τρόποι συνεργασίας. Τι είναι το ETF. Το ETF με λίγα νούμερα είναι ένας οργανισμός που έχει την έδρα του στο Τωρίνο της Ιταλίας. Έχουμε 129 υπαλλήλους και καλύπτουμε 29 χώρες μαζί σας. Ε, ε, έχουμε να μοιραστούμε κάποιες δραστηριότητες του 18. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας που ήρθατε και μας επισκεφθήκατε τον περασμένο Νοέμβριο. Ήταν μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε με τη ε, Κοσλόφσκα Ράντεβιτσι και τον κύριο Κάζα. Επίσης, είμαστε, με χαρά θα υποδεχτούμε οποιονδήποτε θελήσει να μας επισκεφθεί ή έχετε ευθύνε για τις διάφορους γεωγραφικούς οργανισμούς αλλά και τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ευχαρίστως να σας δώσουμε πληροφορίες για τις δραστηριότητες μας σε όλες τις χώρες. Για πέρυσι λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω σε ένα τομέα ε, προβληματισμού που ξεκινήσαμε, το μέλλον δηλαδή να δούμε πώς οι δημόσιες αρχές θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη μετάβαση προς τις νέες δεξιότητες. Ποιος είναι ο ρόλος του δημόσιου τομέα, πώς, τις φέρνουν, πώς φέρνουν τη μεταρρύθμιση στην κατάρτιση και στην παιδεία, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα μέσα που υπάρχουν στις αγορές εργασίας και επίσης αντικατοπτρίζοντας τους διαφορετικούς βαθμούς οριμότητας των αγορών εργασίας εκεί όπου εργαζόμαστε. Το 2019 είναι η 25η μας επέτειος, κλείνουμε τα 25 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε ε, προσβλέποντας το μέλλον και όχι αναπολώντας το παρελθόν. Θα θέλαμε να κάνουμε μια μικρή σύντομη γιορτή στην 1η Νοεμβρίου μαζί με το Διοικητικό μας Συμβούλιο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να γιορτάσουμε αυτήν την επέτειο και να μοιραστούμε μαζί σας κάποια ε, ε, ε στρατηγικές μας για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν τη στρατηγική του ETF 2027. Θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Πέρυσι Προσπαθήσαμε και αναπτύξαμε αυτή τη στρατηγική, εξετάζοντας εξωτερικούς αξιολογητές που μας λένε τι κάνουμε καλά, εξετάζοντας τι επιθυμούν οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και εξετάζοντας πώς αναπτύσσονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπό την καθοδήγηση της DG απασχόλησης, της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, που είναι ε, ε, στο διοικητικό μας συμβούλιο. Επίσης ε, έχουμε τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχει διορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Edith Μπάουερ, Αλεχάνδρο Θέρκας και Φρανσουά Μιζιέ, που είναι οι εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της νέας μας στρατηγικής. ποια είναι αυτή η νέα στρατηγική λοιπόν. Κάναμε μια ανάλυση για το τι συμβαίνει, τι ε, οδηγεί στις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και των δεξιοτήτων και βλέπουμε ότι η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου, η ανάπτυξη δηλαδή δεξιοτήτων αποτελεί ε, μεγάλη προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές δράσεις σε αυτές τις χώρες και για το διάλογο και για την οικονομική βοήθεια. Ε, ε, υπάρχει μεγάλη αλλαγή στα ε, συστήματα τα εκπαιδευτικά και στα συστήματα κατάρτισης. Υπάρχει μεγαλύτερη επαφή ανάμεσα στην παιδεία και την κατάρτιση, περισσότερη συνεργασία με εταίρους που μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματική αποκατάσταση, διαφορετικούς τρόπους μάθησης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην διαβίου ε, μάθηση. Αυτά όλα αντικατοπτρίζονται στο προβληματισμό του Διοικητικού μας Συμβουλίου που συνεδρίασε πριν το καλοκαίρι. Θέλουμε να δούμε ε, εδώ λοιπόν πώς είναι οι δεξιότητες, η παιδεία ε, και Επίσης, ε, να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές της αγοράς απασχόλησης, την ένταξη, τη διαφοροποίηση όσον αφορά τις προσφορές που έχουμε και όλα αυτά να ενταχθούν στις ε, προσεγγίσεις διαβίου μάθησης ε, Να περάσουμε δηλαδή από τις δεξιότητες στην ε, συνεχιζόμενη μάθηση, να μάθουμε από την εμπειρία για το τι σημαίνει στα κράτη-μέλη μας και πώς αυτά μπορούν να μεταφερθούν στις χώρες εταίρους με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Και όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα hub, σε ένα κόμβο γνώσης που θα μπορούν να χρησιμοποιούν και οι Ευρωπαίοι αρμόδιοι για τη λήψη των αποφάσεων. Αυτή είναι η εμπειρία που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, αν θέλετε και αν ενδιαφέρεστε, για τους τομείς συνεργασίας με τις χώρες εταίρους. Τώρα, πώς αναπτύσσουμε και πώς εκτελούμε αυτές τις στρατηγικές είναι μέσω στρατηγικών εταίρων, Έχουμε την οικογένεια του ΟΗΕ, ε, την Σουνέσκο και διάφορους εθνεί ε, οργανισμούς και ακολουθούμε διαφοροποιημένη προσέγγιση, δηλαδή προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας στις ανάγκες της εκάστοτε ε, χώρας. Υπό αυτή την ε, ομπρέλα βλέπουμε τρεις τομείς εργασίας. Έχουμε δηλαδή τις κατάλληλες ε, δεξιότητες και προβλέψεις. Ε, με αυτούς, εδώ συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ακούσατε μόλις το διευθυντή του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες που είναι κοινέ και ενδιαφέρον. Έχουμε δηλαδή δυνατότητα να μοιραστούμε τις γνώσεις μας και να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους εκεί. Βλέπουμε το θέμα ανάπτυξης και κύρωσης, ανάπτυξη των, δηλω... των δεξιοτήτων, δηλαδή και επικύρωση αυτών και ο τρίτο άξονας είναι η απόδοση, τα συστήματα ποιότητας και πολιτικές σε κάθε χώρα. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ο κ. Ζόρντι Καρέλ, της ΕΛΑ του νέου μέλους της οικογένειας σας. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, αισθάνομαι και εγώ ως ε, νέος. Πρώτα απ' όλα γιατί η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι ακριβώς μια νέα υπηρεσία και όπως ξέρετε, επειδή ακριβώς ε, βοηθήσατε κι εσείς ε, να οικοδομηθεί η υπηρεσία μας και ο οργανισμός δημοσιεύτηκε μόλις τον Ιούλιο και οπότε είμαστε σαν ένα νεογέννητο και δεν είμαι ο πραγματικός ε, διευθυντής, είμαι ε, ασκώ καθήκοντα διευθυντού καθώς ε, τους πρώτους μήνες καθώς δεν έχει συσταθεί η υπηρεσία ανετέθη στην Κομισιόν την στήσει οπότε εγώ μαζί με κάποιους συναδέλφους μου εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση Μαζί με τους άλλους διευθυντές των υπηρεσιών θα εξηγήσω και εγώ λίγο σύντομα το σκεπτικό της ε, αρχής αυτής ε, που νομίζω είναι κάτι το χρήσιμο και ε, επίση επειδή έχω και πολύ λιγότερα πράγματα να σας πω ως δραστηριότητες γιατί όπως είπα μόλις 31 Ιουλίου συστάθηκε η αρχή αυτή. Να σας υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε την πρόταση αυτή το 2017. Η πρόταση ήταν μια πρόταση η οποία είχε κατατεθεί το 2018. Νομίζω σε χρόνο ρεκόρ Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συμφώνησαν στον κανονισμό πριν λήξει η προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Αρκετά μεγάλη επιτυχία. Ο κ. Λένατς ήταν ο εισηγητής ε, τότε της πρότασης αυτής και νομίζω είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική προσέγγιση μαζί με την Προεδρία της ε, Ρουμανίας και άρα υπάρχει τώρα αυτή η πρόταση. Τι βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι πράγματι αν δούμε τους αριθμούς η αρχή αυτή θα είναι στην υπηρεσία 17 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που ζουν και εργάζονται σε μια χώρα άλλη από την χώρα προέλευσης τους βεβαίως. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τα πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους ε, εργαζόμενους που είναι αποσπασμένοι κάθε χρόνο. Οπότε μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη αυτή η αρχή. Γιατί προτάθηκε αυτή η αρχή, γιατί η Κομισιόν, ε, όχι μόνο της βεβαίω, γιατί η Συμβούλιο και η Κοινοβούλιο αντέδρασαν γρήγορα, ε, θεώρησε ότι υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ξεκινώντας ε, από το ότι η νομοθεσία είναι ήδη επίκαιρη, όπως ξέρετε. Η Κομισιόν έχει ήδη ενημερώσει την σχετική νομοθεσία, ειδικά όσον αφορά τις αποσπάσεις. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι το σημαντικό είναι η επιβολή αυτών των κανόνων και η επιβολή αυτή είναι κάτι το περίπλοκο όταν μιλάμε για διασυνοριακές ε, καταστάσεις. Βεβαίως οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας έχουν πλήρη αρμοδιότητα στο εσωτερικό της ε, χώρας τους, δεν χρειάζονται στήριξη από το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όταν πρέπει να συνεργαστούν διασυνοριακά μπορεί να βοηθήσει ο φορέας μας. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, η ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή των κανόνων. Το δεύτερο είναι η διοικητική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών φορέων. Δεν μιλάμε μόνο για την εκθεώρηση εργασίας, αλλά για την κοινωνική ασφάλιση και τα σχετικά. Αυτά υπάρχουν ήδη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα, αλλά δεν επαρκούν. Θεωρούσαμε ότι έπρεπε να δοθεί μια όθηση σε αυτήν την συνεργασία. Αυτή ήταν η δεύτερη πρόκληση η τρίτη αφορά την πληροφόρηση και για τους εργαζόμενους που θέλουν να μετακινηθούν και για τις επιχειρήσεις που θέλουν να απασχολήσουν διασυνοριακά. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Το θέμα είναι ότι κάποιες φορές οι πληροφορίες αυτές είναι διασπαρμένες και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Και εδώ πέρα λοιπόν θεωρούμε ότι η αρχή αυτή έχει μια προστιθέμενη αξία και η τελευταία πρόκληση που είδαμε ήταν ότι υπήρχε ένας κατακαιρματισμός στην προσέγγιση όλου αυτού του τομέα. Έχουμε λοιπόν κράτη, στα κράτη-μέλη άτομα τα οποία είναι ειδικά στην απόσπαση αλλά όχι στην κοινωνική ασφάλιση. Άτομα τα οποία είναι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση αλλά όχι στην ελεύθερη μετακίνηση κτλ. Οπότε θεωρήσαμε ότι ένας φορέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ε, συνένωνε την εμπειρία που υπάρχει σε αυτούς τους ε, τομείς θα ήταν κάτι το σημαντικό γι' αυτό στην πρότασή μας ε, όπως ακριβώς την ενέκρινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η αρχή έχει τέσσερις σκοπούς. Η πρώτη, δεν θα σας προξενήσει η έκπληξη, είναι να διευκολύνει πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δεύτερον, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών διοικήσεων. Το τρίτο το οποίο είναι δύσκολο θα έλεγα και οι συζητήσεις ε, μεταξύ των ομοθετών κατέδειξαν την δυσκολία είναι να μεσολαβήσει σε διαφωνίες μεταξύ εθνικών αρχών και βεβαίως ε, να στηρίξει την ε, συνεργασία στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Ε, λοιπόν, αυτοί είναι οι στόχοι οι οποίοι μεταφράζονται σε συγκεκριμένα καθήκοντα αφενός. Έχουμε 7 καθήκοντα τα οποία μας ανέθεσαν. Το πρώτο είναι η πληροφόρηση. Δηλαδή, θα πρέπει να στηρίξουμε τις αρχές ε, στις ε, σχετικές ε, πληροφορίες που αφορούν όλους τους τομείς της ε, κινητικότητας. Να συνεργαστούμε επίσης ταυτόχρονα με τον ενιαίο ψηφιακό κόμβο και να υπάρξει η διαχείριση του δικτύου URES το οποίο ακριβώς φέρνει, έχει όλες αυτές τις πληροφορίες των εθνικών αρχών. Το δεύτερο αφορά την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διοικήσεων, δηλαδή όχι πληροφόρηση του κοινού, αλλά ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών διοικήσεων και εδώ πέρα υπάρχει μια καινοτομία σε σχέση με άλλες υπηρεσίες, ειδικά αυτές οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, που είναι η δημιουργία ακριβώς αυτών των εθνικών συνδέσμων. Δηλαδή αξιωματούχοι αποσπασμένοι από τα κράτη-μέλη που θα έχουν ως καθήκον να λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των εθνικών διοικήσεων θεωρώντας ότι έχοντας αυτούς 27-28 ε, ταυτόχρονα ε, στο ίδιο γραφείο σε καθημερινή επαφή και σε καθημερινή επαφή με την εθνική διοίκηση οι ε, αρμόδιες διοικήσεις ε, θα έχουν καλύτερη επικοινωνία. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της νέας αρχής. Το τρίτο αφορά τον συντονισμό και στήριξη κοινών επιθεωρήσεων γιατί συχνά δεν είναι δυνατό να γίνουν επιθεωρήσεις εργασίας σε ένα κράτος μέλος γιατί υπάρχει διασυνοριακό στοιχείο που θα πρέπει να είναι είτε κοινές ε, από την χώρα που αποσταίνει και λαμβάνει εργαζόμενους ή συντονισμένες, δηλαδή να τις κάνει κάθε εθνική διοίκηση ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης. Το τέταρτο και αυτό είναι πιο παρόμοιο με τις παραδοσιακές υπηρεσίες εδώ γύρω από αυτό το τραπέζι είναι η ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου στον τομέα της κινητικότητας, ένα πέμπτο καθήκον για την δημιουργία ικανοτήτων σε εθνικές διοικήσεις μέσω της παροχής εκπαίδευσης του προσωπικού και βελτίωσης της δυνατότητας συνεργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον. Το έκτο είναι να δούμε τις δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, οπότε δεν θα χαθεί αυτή η πλατφόρμα, αντιθέτως θα ενταχθεί ε, στην αρχή μας και τέλος ε, μια καινοτομία να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ε, διαιτησίας μεταξύ των διοικήσεων σε περίπτωση διαφωνίας. Οπότε αυτά είναι τα καθήκοντα που έχουμε, νομίζω είναι ξεκάθαρο. αφορά την κινητικότητα θα καλύπτουμε όλους τους τομείς, είτε μιλάμε για την ελεύθερη μετακίνηση, μηχανισμούς ε, και συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, απόσπαση και θα καλύπτουμε όλους τους κλάδους. Αλλά βεβαίως ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον τομέα των οδικών μεταφορών λόγω της φύσεώς του και της φύσεως του η οποία σημαίνει μεγάλη κινητικότητα. Οπότε θα καλύψουμε όλους τους κλάδους, όπως είπα, με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς οδικές μεταφορές. Οπότε η αρχή αυτή δεν γεννήθηκε εν κενό. Θα έχει πολύ στενή συνεργασία με την πλατφόρμα που υπάρχει για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επίσης με το δίκτυο EURES, μια που το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού θα ενταχθεί στην αρχή αυτή επίσης και βεβαίως θα υπάρχουν όλα αυτά τα δίκτυα για τις αποσπάσεις και τα λοιπά και θεωρούμε ότι με το να συνανωθούν όλα αυτά τα δίκτυα και ομάδες θα έχουμε μεγαλύτερες συνεργίες και θα ενισχύσουμε έτσι, την αποτελεσματική λειτουργία όλων των εργαλείων που είναι στη διάθεσή μας και βεβαίως θα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς και πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά κύριο λόγο με τις φυστάμενες υπηρεσίες και το Eurojust και τη Europol. Μιλάμε για τις εθνικές επιθεωρήσεις ε, βεβαίως ε, και έχουμε και ζητήματα που αφορούν την Eurojust και τη Europol. Λοιπόν, ποια θα είναι η διοικητική δομή τώρα της αρχής αυτής. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει ένας εκτελεστικός διευθυντής και οι διαδικασίες για ε, τον διορισμό της θα ξεκινήσουν αμέσως. Μετά θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο αυτό βεβαίως θα υπάρχουν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, ε, της Κομισιόν, ένας ε, ειδικό που θα ορίσει το Κοινοβούλιο και εκπρόσωποι και των εργαζομένων και των εργοδοτών και βεβαίως ε, δεν θα περιορίζεται μόνο σε ευρωπαϊκές ε, χώρες αλλά θα επεκταθεί και σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εφαρμόζουν τους κανόνες όπως Ισλανδία, Ελβετία, Νορβηγία κτλ. Πέρα από αυτό λοιπόν θα υπάρχει και η ομάδα των ενδιαφερομένων μερών που θα εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί εταίροι, θα παίζει έναν συμβουλευτικό ρόλο και θα γνωμοδοτεί κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μια σημαντική απόφαση. Θα ζητείτε η γνώμη των ε, ομάδων συμμετεχόντων. Ερχόμαστε τώρα στα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα χρόνο διάγραμμα, θα υπάρξει μια αρχική φάση 5 ετών, μόλις ξεκινήσαμε. Σταδιακά η αρχή θα αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία αυτή τη στιγμή κάνει η Κομισιόν, αναφέρομαι στη EURES, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αδήλωτη Εργασία και αυτό θα γίνει με τρόπο προοδευτικό, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως το πώς το ε, προσωπικό θα προσλαμβάνεται και έχοντας ε, πάντα κατά νου την συνέχεια της λειτουργίας. Δεν θέλουμε να διαταράξουμε ε, υπηρεσίες που παρέχονται, ήδη όπως η EURES, η πλατφόρμα, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να φροντίσουμε να μην υπάρχει κάποια διακοπή της λειτουργίας. Αντιθέτως όλα αυτά να μεταφερθούν. Ε, οπότε στο τέλος της πενταετούς ε, περίοδου όταν η αρχή αυτή θα έχει φτάσει μια κανονική λειτουργία θα έχει γύρω στα 140 άτομα προσωπικό και έναν προπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως ε, φέτος, μια που υπάρχουν μόνο 4-5 μήνες και πάρα πολύ μικρές δραστηριότητες, ο προπολογισμός είναι πολύ πιο μικρός, είναι 2,1 εκατομμύρια. Θα αυξάνεται βεβαίως. Οπότε, πού βρισκόμαστε σήμερα. Όπως είπα, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εργάζεται ένεργα για να στηρίξει την δημιουργία αυτής της αρχής. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την φάση των προσλήψεων για να φτάσουμε σε 20 άτομα προσωπικό μέχρι το τέλος του έτους και 60 ε, άτομα μέχρι το 2020. Βλέπετε ότι έχουμε φιλόδοξους στόχους, ειδικά αν σκεφτείτε την ε, δυσκίνητη διαδικασία προσλήψεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον επόμενο μήνα 16 και 17 Οκτωβρίου και εκεί πέρα βεβαίως θα έχουμε τους εκπροσώπους των κρατών μελών, των συνδικάτων, του Κοινοβουλίου, των υπηρεσιών των υπολείπων και πέρα από κάποια πράγματα εσωτερικά, έγκριση του κανονισμού κτλ. Ε, θα έχουν δύο ουσιαστικά καθήκοντα. Το ένα θα είναι να εγκριθεί η δημοσίευση της περιγραφής του ε, αντικειμένου εργασίας ε, της Διευθύντριας και το δεύτερο θα είναι να υπάρξει μια συζήτηση για το πρόγραμμα εργασίας για το 2020. Αναφέρθηκα στα 7 καθήκοντα. Είναι προφανές ότι τα 7 καθήκοντα δεν θα αρχίσουν να εκτελούνται από την πρώτη στιγμή πλήρως, δεν υπάρχουν πόροι, οπότε θα πρέπει να ληφθεί μια στρατηγική απόφαση περί προτεραιοτήτων. Ποια από τα 7 καθήκοντα θα είναι τα 2-3 που θα είναι τα πιο σημαντικά για να μας αποσχολήσουν αμέσως. Βεβαίως, ε, ως ε, ε, προσωρινός διευθυντής δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση του ΔΣ. Και υπάρχει μια συζήτηση. Έχουμε προβλέψει λοιπόν ένα ΔΣ αρχές Δεκεμβρίου και να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε το επόμενο έτος. Λοιπόν, Αυτά είναι τα βασικά. Βεβαίω κάτι το οποίο όλοι γνωρίζετε είναι ότι η έδρα θα είναι στην Μπαρατισλάβα και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές της ε, Σλοβακίας για να τις βοηθήσουμε έτσι ώστε το κτίριο που υπάρχει ήδη να ε, συμμαζευτεί για να μπορέσει να μετακινηθεί εκεί το προσωπικό το συντομότερο δυνατόν. Οπότε Καταλήγω λέγοντας ότι γνωρίζουμε το ότι η σύσταση της αρχής αυτής έχει δημιουργήσει πολλές προσδοκίες και θα παραμείνει ψηλά στην πολιτική ατζέντα και για τη νέα κομισιόν. Όπως ξέρετε η νέα πρόεδρος η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει περιλάβει την εύρυθμη λειτουργία της αρχής μας στην αποστολή του νέα επιτρέπου για την εργασία. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε σωστά, να υπάρχει η στρατηγική κατεύθυνση από το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, για να συνεργαστούμε όλοι έτσι ώστε να είναι επιτυχέ το νέο αυτό εγχείρημα. Ευχαριστώ. Κύριε Κρόλ, κοιτάξτε, επειδή θα είσαστε στην Πατισλάβα, στην χώρα μου, στην πατρίδα μου, σας άφησα να μιλήσετε για τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ρεαλιστικό και ο πραγματικός ο χρόνος που βλέπουμε στην οθόνη, διότι κατά λάθο ξέχασα να σταματήσω το χρονόμετρο. Μόνο τέταρτο ήταν και όχι 25 ο χρόνος για τον οποίο μιλούσατε. Οπότε ερχόμαστε στο πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές ο κ. Ράτκα θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, δουλειά που έχετε κάνει η οποία είναι προσθέμενη αξία και για εμάς αλλά και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις ε, και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο ότι έχουμε πολλούς νέους ε, βουλευτές ε, στην Επιτροπή μας και το οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες από πρώτο χέρι παρατήρησα ε, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας υπάρχει ακόμα αυτή η άβρα του νέου. Χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα. Έχω τώρα δύο συγκεκριμένα πράγματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Πρώτα απ' όλα ο κ. Ζήμπελ αναφέρθηκε στο ότι ο ίδιος θα ήθελε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ε, κατάρτιση, κάτι το οποίο βέβαιως με αφορά ιδιαίτερα γιατί αφενός βλέπω διαφορά προβλήματα, έχουμε περιοχές οποίες ε, δεν θεωρείται η κατάρτιση ισότιμη, ε, δηλαδή δεν υπάρχει και κάτι το επίσημο, απλά κάθε εκεί και δουλεύει στο πλάι και μαθαίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια σε περίοδους κρίση και το άλλο είναι ότι στη Γερμανία μου, στη Γερμανία, στη χώρα μου θεωρείται η κατάρτιση κάτι το οποίο ας πούμε είναι για αυτού που δεν ήταν αρκετά έξυπνοι για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Δεν ισχύει όμω, Αν δείτε ε, χάρη σε πόσες εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις ε, είναι διευθυντής κάποιος ο οποίος ε, είχε κάνει μια τέτοια επιχείρηση. Ο αν δείτε και παραδείγματο χάρη και σε μεγάλες επιχειρήσεις, την Bayer παραδείγματο χάρη στο ΔΣ, τα βιογραφικά των μέλων. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να σας πω, αναφερθήκατε στο ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, πράγματι αυτό ισχύει, αλλά ειδικά στην απόσπαση αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα, ότι έχουμε κράτη τα οποία δεν τηρούν του κανόνε, δηλαδή αν δούμε το πιστοποιητικό 1α ε, υπάρχουν ε, παραδείγματος χάρη α1 βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, γραφειοκρατικά εμπόδια σε Γαλλία, Βέλγιο και Αυστρία όπου έχουμε και αποφάσεις του ΔΕΚ γιατί αγνοούν τα πιστοποιητικά αυτά τα α1 και υπάρχουν και πρόστιμα κτλ. Το θέμα είναι λοιπόν πώς βλέπετε τον ρόλο σας ε, στην μείωση της ε, γραφειοκρατίας για να μπορέσουμε τελικά εντάξει, να εμποδιστεί η κατάχρηση των κοινωνικών παροχών αλλά να μειωθεί και η γραφειοκρατία. Κυρία Μπίσοφ, ε, η ερωτήση σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις παρουσιάσεις σας. Έχουμε 60% νέα μέλη στην Επιτροπή και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο όσον αφορά το σχεδιασμό πολλών από αυτές τις αρχές, από τους οργανισμούς και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Όλοι αναφερθήκατε στους φορείς αλλαγής, ψηφιοποίηση, αλλαγή του κλίματος, μετανάστευση, δημογραφικές αλλαγές. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω τις βασικές προτεραιότητές σας όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα όσον αφορά τους φορείς αλλαγής. Ακούσαμε την παρουσίαση της ΕΛΑ. Είσαστε καινούριος φορέας. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι πολύ σημαντική σημαντικό το έργο Αν θέλουμε να εγγυηθούμε ελεύθερη μετακίνηση και στο μέλλον, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και καλύτερους ελέγχους. Ερώτηση. Για να από τα βασικά θέματα. Ο κύριος Γιούνκερ στην ακρόασή του εδώ είχε αναφερθεί στην εγγύηση της αρχής ίσης αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί μέσα στις προτεραιότητες σας, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ο κ. Πισλάου για το Renew Europe. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε το έργο σας και μελλοντικά προγράμματά σας και τα επιτεύγματά σας. Επανειλημμένα έχω αναφέρει τη σημασία τριών στοιχείων που επηρεάζουν την εργασία σας. Πρώτα απ' όλα να παράγονται τα αναγκαία στοιχεία για το Κοινοβούλιο διαμορφώνει εμπεριστατωμένη πολιτική. Μετά, η προπτική που αναφέρατε για τα μελλοντικά προβλήματα, δημογραφικά προβλήματα, ψηφιοποίηση, να μετανάστευση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Και κάτι άλλο. Η άποψή μας να έχει στο επίκεντρο τον πολίτη. Για το ΕΛΑ πρώτα. Ο νέος οργανισμός. Έχω μία ερώτηση. Είμαι σκιώδης εισηγητής για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Κάποιοι έλεγαν ότι ο φορέας σας θα είναι η λύση για την εφαρμογή, για την υλοποίηση της πολιτικής. Συμφωνώ ότι η συνεργασία είναι καλή, αλλά η ψηφιοποίηση των κοινωνικών συστημάτων ασφαλείας είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα υπάρξει συντονισμός των διαφόρων φορέων. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο τελικά να μην επιβαρύνει τους πολίτες αλλά τον φορέα για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Αναφέρθηκαν οι διάφορες εκθέσεις για προβλέψεις, για τα μελλοντικά προβλήματα και τα επιτεύγματα. Χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παιδεία. Ξέρουμε τα όρια που επιτάσσουν οι συνθήκες. Η θεωρητική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Πώς ενώνονται σε μια κοινή προσέγγιση Αυτές οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους. Η κυρία Μαρή Πίτερ Χάνσεν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Πολύ σημαντικό το έργο σας για την κοινωνική Ευρώπη. Σαν νέα Ευρωβουλευτής ενδιαφέρθηκα πολύ για αυτά που άκουσα. Έχω ερώτηση όσον αφορά τη διαφάνεια για την αμοιβή των δύο φίλων. Κυρία Μενέντες Βαλτές, λεπτομέρειες θα ήθελα. Η έρευνά σας τι έδειξε και βάσει της εκθέσεως που ετοιμάσατε για τις αμοιβέ στις τέσσερις χώρες. Ποια είναι η άποψή σας. Ποια νομοθεσία λειτουργεί. Πώς μπορεί να μειωθεί η διαφορά των αμοιβών ε, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. ID κυρία Ζαμέ που δεν είναι εδώ άλλος από το ID όχι η κυρία Ραφάλσκα για το ECR Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας και για την εδώ παρουσία σας και που αναφερθήκατε στα προβλήματα Έχουμε οργανισμούς που επιμακρών λειτουργούν. Κάποιοι από τους οργανισμούς έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 40 χρόνια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τι κάνετε. Κυρίως διότι υπάρχουν πολλοί νέοι ευρωβουλευτές και ήταν καλές εξηγήσεις. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και για τις εξηγήσεις που δώσατε. Έχουμε έναν κοινό παρονομαστή στα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα. Ποιο είναι ο παρονομαστή, η γύρανση του πληθυσμού που λαμβάνει η χώρα παντού. Είναι θέμα που αναφέρατε περισσότεροι από εσά. Άλλο θέμα είναι η ψηφιοποίηση, κοινό στοιχείο στι παρουσιάσει σα. Και οι νέε απειλέ όσον αφορά τι θέσει εργασία. Προβλήματα που προκύπτουν από τη γύρανση του πληθυσμού αλλά και από τη μετανάστευση. Μία γενική ερώτηση που απευθύνω σε όλους σε όλους τους οργανισμούς. Πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από τα αποτελέσματα της δουλειάς που κάνετε, οι εκθέσεις σας, οι στατηγικές σας χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται από εκείνους που διαμορφώνουν την πολιτική. Ακούσαμε και μακροσκελή παρουσίαση που αφορούσε το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας και οι προλαλήσαντες αναφερθήκαν στις διάφορες προσδοκίες που υπάρχουν όσον αφορά το ELA. Θεωρείται σημαντική η προστασία των εργαζομένων και των μεταναστών εργαζομένων. Υπάρχουν νομοθετικές αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί και αφορούν την ίση αμοιβή. Ε, μιλώ εκπροσωπώντας την Πολωνία που έχει το μεγαλύτερο αριθμό αποσπασμένων εργαζομένων σε άλλες χώρες. Περίπου μισό εκατομμύριο αποσπασμένους εργαζομένους έχουμε. Ξέρουμε ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι ακόμα μεγαλύτερη ομάδα από τους αποσπασμένους εργαζομένους. Είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα στην εκμετάλλευση ίσως να μην γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία εργάζονται. Ίσως να έχουν συμβάσεις μηδενικών ωρών, ορισμένου χρόνου. Έχουμε εθνικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με το σεβασμό του εργασιακού δικαίου. Σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξει αυτός ο σεβασμός. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχω και άλλη ερώτηση. για την αρχή για την υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασία. Αν συλλέγονται στοιχεία από εργαζομένους που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας που πάσχουν από κατάθλιψη φερρυπίν. Ίσως αυτό να συνδέεται με δημογραφικά προβλήματα, με τη γύρανση του πληθυσμού και με τους ανθρώπους που χάνουν την υγεία τους. Αυτό αντικατοπτρίζει στις υγείες σα, εκθέσεις σας. Διότι ε, στις εκθέσεις αναφέρεται ότι πρέπει να εργαζόμεθα όλο και περισσότερο. Ποια είναι τα όρια των εργαζομένων. που να περισσότερα ή όχι όσο γυράσκουν. Ευχαριστώ. Ο κ. Βιόμψεν για την Γκουε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε όλους σας που ήρθατε, λέει ο κ. Βιόμψεν και τις προσπάθειές σας. Όπως και άλλοι, θα εστιαστώ επί του ΕΛΕ, που είναι ο νέος μαθητής του ΣΥΠΗΝ. Θα ξεκινήσω από κάτι που είναι ε, περισσότερο σχόλιο από ερώτηση. Σύντομα, θα έχουμε το διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΑ που για πρώτη φορά θα συνεδριάσει. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικότατο να εξασφαλίσουμε την παρουσίαση των συνδικάτων. Είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑ στο μέλλον. Θα ήθελα ξεκινήσω λοιπόν υπογραμμίζοντας ότι ελπίζω πραγματικά ότι η ρήτρα περιεμπιστευτικότητας δεν θα χρησιμοποιηθεί για να εξαιρεθούν οι κοινωνικοί εταίροι, να αποκλειστούν οι κοινωνικοί εταίροι. Υποθέτω ότι συμφωνείτε με αυτό αλλά είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε παρόλα αυτά. Μία ερώτηση έχω για σας, κύριε Τζόρντι Κοέλ Γκατόρ, εάν προφέρω σωστά το όνομά σας, ο ΕΛΑ πώς θα εφαρμόσει συγκεκριμένα τις διατάξεις περί κοινωνικών εταίρων του άρθρου 8 του κανονισμού του ΕΛΑ. Δηλαδή ότι οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να πιστήσουν την προσοχή του ΕΛΑ σε διάφορα προβλήματα, ούτω ώστε να ξεκινήσουν έλεγχοι μεμονωμένοι ή από κοινού. Θα ήθελα απάντηση σε αυτό, διότι είναι κρίσιμο στοιχείο για να λειτουργεί εύρυθμα ο ΕΛΑ. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε για να μας διαφωτίσετε για το έξοχο έργο που επιτελείτε. Thank Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Ήδη έχουμε υποβάλει και αρκετά ονόματα. Ε, έχω μάλλον καταγράψει τα ονόματα όσων θέλουν να θέσουν ερωτήσεις στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων και θα δώσω το λόγο τώρα στους προσκεκλημένους μας και επειδή ε, οι περισσότεροι ερωτήσεις αφορούσαν το ΕΛΑ θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κορέλ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο στην πρώτη μου εισήγηση. Νόμιζα πως επειδή ήμουν ε, νεοφερμένος, χρειαζόταν κάποιες εξηγήσεις για το τι κάνουμε. θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα υπόψη μας ποιος είναι ο ρόλος του ΕΛΑ σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο ρόλος του ΕΛΑ αφορά την ε, επιβολή και την εφαρμογή και διευκόλυνση της επιβολής. Δεν είναι ο ρόλος μας να φτιάξουμε νέα νομοθεσία και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Όπως γνωρίζετε, η, η τελευταία τροποποίηση της σχετικής οδηγίας προβλέπει αυτή την αρχή και το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην πρώτη του ομιλία ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου. Αυτή η οδηγία τώρα λοιπόν έχει εγκριθεί, δεν έχει αρχίσει ακόμα να ισχύει, αλλά ο ρόλος του ΕΛΑ Πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο ρόλος της Κομισιόν ως ε, θεματοφύλακα της συνθήκης, γιατί εκείνη θα πρέπει να να δει και να μεταφράσει, ε, να ελέγξει κατά πόσο τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την ε, νομοθεσία στην εθνική νομοθεσία. Αυτός είναι ο ρόλος της Κομισιόν και όταν εμείς όμως μπορούμε να συνεργαστούμε και να δούμε, όταν μάλλον διαπιστώσουμε μία εφαρμογή της νομοθεσίας, ε, ας πούμε όταν υπάρχει μια εταιρεία βιτρίνα και τα λοιπά, ε, να ε, συνεργαστούμε και να ενημερώσουμε. Και έτσι έρχομαι στην ερώτηση του κύριου Ράτκε για την άρση της γραφειοκρατίας, για την κατάρριση της γραφειοκρατίας. Τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Όντως κάποιες φορές οι κανόνες είναι οι κατάλληλοι, αλλά κάποιες φορές η εφαρμογή τους επιτόπου δεν λειτουργεί ορθά. Και γι' αυτό το λόγο η συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς διοικητικούς μηχανισμούς είναι πολύ σημαντική. Κάποιες φορές η συνεργασία είναι πολύ καλή, αλλά άλλες όχι. Πρέπει δηλαδή συχνά να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμά και τις εθνικές διοικήσεις. Αυτό για να γίνει χρειάζονται να εξασφαλίσουμε τους πραγματικούς κανόνες, δηλαδή αυτούς που χρησιμοποιούνται και ισχύουν και κατά πόσο είναι προσαρμοσμένοι. Άρα λοιπόν πρώτα θέλουμε να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο και όταν θα έχει αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο και θα έχει μπει σε ισχύ, θα έχει τεθεί σε ισχύ, τότε ε, θα δούμε ποια θα είναι η νέα ε, κουλτούρα συνεργασίας. Ε, να πείσουμε εμείς θα πρέπει ότι υπάρχουν τρόποι συνεργασίας πέρα από την τυπική. Εκεί έχουμε μετά να παίξουμε σημαντικό ρόλο. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο και ειδικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν σαφείς και ε, αποφασιστικές ε, υποδείξεις ε, στους NLO για να συνεργαστούν μεταξύ τους. Επίσης, εσείς αναφερθήκατε στα συστήματα πληροφορικής. Ξέρετε βέβαια ότι εργαζόμαστε εντατικά με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή και για το στήσιμο του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό θα είναι σπουδαία αλλαγή. Ένα είναι μεγάλο project και δύσκολο 15.000 ε, ε, θεσμοί κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά περίπλοκο ε, εγχείρημα, αλλά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε μπει τώρα στην τελική φάση και αυτό θα κάνει τη ζωή των πολιτών πολύ, πολύ ευκολότερη. Αυτό είναι βέβαιο. Βέβαια, είμαστε στη μέση της ε, Κομισιόν. Εγώ μόλις ε, ορίστηκα, διορίστηκα διευθυντής. Υπάρχει ένα project όμως που έχει αναφερθεί και προηγουμένως για το Ευρωπαϊκό Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό θα αποτελέσει σπουδαία αλλαγή για τους ε, Ε, και βεβαίως ε, θα ε, είναι μεγάλη αλλαγή όταν θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Κάτι ακόμα, ρωτήσατε για τον αντίκτυπο της δικής μας εργασίας, αλλά αναφερθήκατε Επίσης, αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πείτε εσείς και θα με ρωτήσετε αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργα... μάλλον τι γίνεται με αυτούς που δουλεύουν αποσπασμένοι σε άλλη χώρα της Ένωσης. Υπάρχει σχετική οδηγία που ρυθμίζει την ε, συγκεκριμένη περίπτωση. Η ισότητα ε, ισχύει εκεί ε, ανάμεσα στους υπηκόους και τους μη υπηκόους των ευρωπαϊκών χωρών. Η να, ο ΕΛΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει οδηγία από το 2014 που ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν πως έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό για να ελέγξουν το σωστή εφαρμογή των βασικών αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου και αυτή η οδηγία, όπως είπα, από το 2014 ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν πως υπάρχουν συγκεκριμένα σώματα που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους και είμαι βέβαιος πως η εν λόγω αρχή θα μπορέσει να φέρει αυτά τα σώματα, τα εθνικά σώματα σε συνεργασία. Ε, ελπίζω λοιπόν πως ε, σε λίγα χρόνια ο τότε διευθυντής θα μπορέσει να έρθει ενώπιον της Επιτροπής σας και να σας δείξει με στοιχεία ποιος είναι ο αντίκτυπος και επιρροή της δικής μας εργασίας. Ρόλος των συνδικάτων. Ρόλος των συνδικάτων ρωτήσατε και ρόλος της ETUC που ε, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε ήδη ε, επικοινωνία με την ETUC, έχουμε δύο εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να εξασφαλίσουμε πώς θα δημιουργηθούν οι ομάδες των stakeholders όσο γίνεται πιο σύντομα. Για το άρθρο 8 που είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε όπως και εγώ ότι δεν ήταν το ευκολότερο ε, άρθρο στη διαπραγμάτευσή του. Είχαμε ιδιαίτερα δύσκολες διαπραγματεύσεις εκεί θα έχουμε εδώ να κάνουμε με διαπραγματεύσεις και διαμαρτυρίες ή καταγγελίες από όλους, αλλά κυρίως από τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουν ρόλο να παίξουν οι κοινωνικοί εταίροι στα κράτη-μέλη. Και όσον αφορά την, ε, εργασία, ε, την επιθεώρηση εργασίας, εκεί κάποιες φορές τα ίδια τα, τα, τα συνδικάτα της προβαίνουν σε αυτές τις επιθεωρήσεις, ενώ σε άλλα κράτη όχι υπάρχουν επιθεωρήσεις εργασίας. Θα πρέπει ωστόσο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σεβόμενοι τα διαφορετικά εθνικά συστήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ζίμπελ και μετά ε, ο κύριος Βάλτες. Μάλιστα. Για την ερώτηση του κύριου Χάρκη, συμφωνώ μαζί σας ότι η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να είναι ε, ένα ομαλό μονοπάτι και όσον αφορά την τυποποίηση της κατάρτισης και ε, της δυνατότητας σύγκρισης κράτη-μέλη και εδώ συμφωνώ μαζί σας και αυτό το κάνουμε στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ε, προσφέρουμε τέτοια project. Τελευταία είχαμε ένα με την Μάλτα και ένα με τη Σλοβακία, όπου βοηθήσαμε να ε, ενημερώσουν τις διαδικασίες και τις πολιτικές και αυτό το κάνουμε περισσότερο προσπαθώντας να βοηθήσουμε. Δεν δίνουμε οδηγίες. Ε, θα πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση ανάμεσα στους εθνικούς ε, ενδιαφερόμενους φορείς και μας. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα τώρα και εδώ μπορώ να σας πω μόνο πως η δυνατότητα απασχόλησης είναι πολύ βασική για, τον, για έναν εργοδότη και η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα πρότυπο που πραγματικά εξοπλίζει τους νέους με την δυνατότητα απασχόλησης γιατί έχουν ένα μεγάλη δυνατότητα έτσι να μάθουν πρακτικά και επίσης προέρχομαι από μια εξατία από 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι τρεις ξεκίνησαν από μαθητεία, ως μαθητευόμενοι. Δεν είναι η μόνη βέβαια ε, ε, ε, δεξιότητα. Αργότερα έχουμε φτάσει και στα διδακτορικά. Η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι ανώτατο όριο, δεν είναι πλαφόν. Είναι όμως μία διοχέτευση, ας πούμε, ένα κανάλι από το οποίο μπορεί κανείς να μετακινηθεί πιο εύκολα μετά σε θέση απασχόλησης. Συνδυάζουμε λοιπόν τώρα τη θεωρητική γνώση με την πρακτική γνώση και εδώ πιστεύω πως η επαγγελματική κατάρτιση είναι το πρότυπο που διευκολύνει σε αυτό γιατί πάντοτε συνδυάζει τα θεωρητικά μαθήματα με τις εφαρμοστές μένες ευκαιρίες μάθησης είτε είναι σε επαγγελματικά σχολεία είτε είναι στην ε, μαθητεία σε κάποια ε, εταιρεία κοντά στον εργοδότη δηλαδή. Επίσης, τα σενάρια που μοιράστηκα μαζί σας νωρίτερα, ένα από αυτά συμπεριλαμβάνει την ιδέα της επέκτασης αυτής, της, αυτού του συνδυασμού στην ανώτατη εκπαίδευση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 κυρία Ράφακ, ε, οι ερωτήσει που έκανε σε σχέση με τον αντίκτυπο του και το κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα, ναι, από την εμπειρία μου στον ιδιωτικό τομέα, εγώ να σας πω ότι χρησιμοποίησα τα αποτελέσματα του ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη δουλειά μου, γιατί υπάρχουν ενημερωτικά δελτία εξαιρετικά για κάθε χώρα, βοηθάνε να αξιολογήσουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα επαγγελματική κατάρτισης σε κάθε χώρα και πώς εμείς ως εργοδότες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα συστήματα συστήματα και να υποφεληθούμε από αυτά. Βέβαια αυτό δεν είναι επιστημονικές αποδείξεις, το ξέρω. Ε, ε, ε, ωστόσο, είδατε και μια από τις διαφάνειες που σας παρουσίασα σύντομα, και λέω κάποια νούμερα, ας πούμε, οι δημοσιεύσεις έχουμε 345 ε, χιλιάδες φορές ε, κατέβασαν αυτά τα στοιχεία χρήστες. Έχουμε επισκέψεις στο Europass, έχει φτάσει στις 16, τα 16 εκατομμύρια επισκέψεις. Ε, έχουμε διάφορα έγγραφα και δημοσιεύσεις που φτάνουμε ε, όπου αναφερόμαστε σε επιστημονικές ε, δημοσιεύσεις ε, πάρα πολλές φορές και θέλω να επενέσω όλο μου το επιτελείο. Είναι εξαιρετική όλη στη Θεσσαλονίκη και φτάνουν ε, σε τόσο πολύ κόσμο. Νομίζω λοιπόν πως δημιουργούμε, πως, πως ακουγόμαστε αρκετά. Νομίζω πως αυτές ήταν οι ερωτήσεις που μου απευθύνατε εμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και κυρία Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις ε, ε, διαφόρων βουλευτών για το τι κάνουμε για την ίση αμοιβή ένα θέμα ισότητας των φύλων είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Του χρόνου θα εφαρμόσουμε τον επόμενο γύρο ε, της μελέτης για τις ε, συνθήκες εργασίας. Θα έχουμε πολλά νέα στοιχεία όσον αφορά το ωράριο εργασίας, την ευελιξία, τους μισθούς, ε, ε, την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και ιδιωτικής ζωής, ε, θα έχουμε ένα σωρό νέα, και φρέσκα στοιχεία. Επίσης είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι εμείς ρωτάμε τον κόσμο για το πόσες ώρες εργάζονται και πόσες θα ήθελαν να εργάζονται. Και επίσης πόσο, πόσα μέλη εξαρ, έχουν ε, εξαρτώμενους ε, και γενικά βλέπουμε πως η τάση είναι προσμείωση των όρων απασχόλησης. Για την επόμενη πολιετή μας έρευνα έχουμε στοιχεία που θα συνδυάζουν ε, την έρευνα των οικοκυριών με την έρευνα ε, των συνθηκών εργασίας. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ε, για την ισορροπία όλων αυτών εάν δεν ρωτήσουμε ε, τους ανθρώπους που μένουν στο σπίτι. Τα πράγματα λοιπόν μπορείς να τα δεις έτσι καλύτερα. Δεν μπορείς να ρωτάς μόνο εργαζόμενους. Αλλά πρέπει να ε, έρθει σε επαφή και με τους μη εργαζόμενους για να λέξει στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ρόλο τους, με την κατανομή των καθηκόντων κτλ. Για την διαφάνεια στους μισθούς. Η κυρία Πέτρε Χάνσεν Έθιξε αυτό το ερώτημα. Δημοσιεύουμε έκθεση για την εφαρμογή των συστάσεων στα κράτη-μέλη. Βασικά υπάρχουν δύο μοντέλα ε, χωρών. Υπάρχουν χώρες που είναι πιο απαιτητικέ και που οι αναφορές περί των εταιριών είναι πιο εκτεταμένες και άλλες όπου ε, τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα και πρέπει να δημοσιεύουμε κάποιες ε, πολύ βασικές πληροφορίες. Όσο πιο επαιτητικός είσαι, τόσο πιο πλούσιες πληροφορίες ε, παίρνει, αλλά έχεις λιγότερο, χαμηλότερο ε, επίπεδο ανταπόκριση. Εάν ζητά λίγα πράγματα, ε, σου απαντάνε περισσότεροι, αλλά δεν έχεις αρκετές πληροφορίες, δεν βγάζει νόημα. Εδώ θα το δουλέψουμε περισσότερο και θα επανέλθουμε μόλις ε, θα ξέρουμε ποιες χώρες το έχουν εφαρμόσει αυτό για να δούμε ποιο είναι είναι η επιβάρυνση. Τώρα, για τις εργασιακές σχέσεις μπορώ να μιλάω για όση ώρα θέλετε γι' αυτό. Δεν έχουμε όμως χρόνο να πω όμως ε, στις δύο θεματικές προσεγγίσεις ε, που προτείνουμε για τον επόμενο πολιετή κύκλο. Το ένα είναι για την κοινωνική συνοχή και τη σύγκληση κοινωνική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνοδεύουμε όλη τη διαδικασία που συνδέεται με το εξάμεινο κτλ. Αλλά και να δούμε πως εντός των ε, κρατών μελών οι κοινωνίες έρχονται πιο κοντά και εκτός και μεταξύ δηλαδή κρατών μελών και εδώ πάλι έχουμε Έχουμε να κάνουμε με προβλήματα με τις επερχόμενες ε, αναδιαρθρώσεις. Πρέπει να δούμε δηλαδή προσεκτικά κάποια στοιχεία. Έχουμε κάποιες ε, δημοσιεύσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να δούμε δηλαδή τα θετικά όσον αφορά την κοινωνική ε, προστασία των εργαζομένων. Τέλος, και ίσως σε σχέση με ένα θέμα που αφορά το πώς ε, ε, παρακολουθούμε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αξιολόγηση, ποια είναι η παρακολούθηση. Έχουμε εξωτερικό συνεργάτη, έχουμε ένα σύστημα δικτών, το ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουμένως, έχουμε 273, 273 ευρωπαϊκά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν τα πορίσματα του Eurofind. Ε, έχουμε ε, επίσης χρησιμοποιηθεί βασικός χρήστης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έχουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Είναι φυσιολογικό ότι ο κύριος χρήστης των δικών μας μετρήσεων και πορισμάτων είναι η Κομισιόν. Όμως και αρκετές από τις δικές σας εκθέσεις, σε δικές σας εκθέσεις πρωτοβουλίας έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία του Eurofound. Το ΑΕΛΟ κάνει τέτοιες μελέτες επίσης, το Διεθνής Οργανισμός, το Διεθνές Γραφείο ε, Εργασίας. Και πάλι όμως η Κομισιόν είναι ο βασικός χρήστης. Τώρα, επιστημονικές παραθέσεις που είναι σημαντικός έμεσος δείκτης για μας, γιατί δεν συνδέεται τόσο πολύ με το πόσο ε, χρησιμοποιεί την εργασία μας, αλλά με το πόσο αξιόπιστος είναι. Ε, εδώ πρέπει να δούμε ποιες είναι οι χρήσης αυτών των ε, ε, στοιχείων από τα ε, διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σελατσεκ. Έχετε τον λόγο και να ετοιμάζετε ο κύριος Ωνεσίνη. Ε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τις γενικές ερωτήσεις που αφορούν την συνεισφορά μας και τη στήριξη στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Λίγο πολύ θα έλεγα και αυτό περιλαμβάνεται και στο πολυετές στρατηγικό μας ε, πρόγραμμα οτιδήποτε κάνουμε βασίζεται στα αιτήματα και τις ε, ερωτήσεις ε, που υπάρχουν στα θέματα στον κοινωνικό πυλώνα. Δηλαδή θεωρούμε ότι η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι ανθρώπινο δικαίωμα και αυτή είναι η βάση των όσων κάνουμε. Να αναφέρω τώρα κάποιες προτεραιότητες Νομίζω το ανέφεραν όλοι οι συναδελφοί μου. Ψηφιοποίηση τελειώσαμε μια δραστηριότητα σε τέσσερα σημεία. Ε, με Κάναμε κάποια μελλοντικά σενάρια για το τι θα συμβεί υπό ορισμένε συνθήκε. Παραδείγματο χάρη, αν υπάρξει ύφεση στην οικονομία, εάν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες επενδύσεις για την ψηφιοποίηση, ή για την διαβίου κατάρτιση. Οπότε τώρα έχουμε μια αρκετά καλή βάση για να προετοιμάσουμε μια γενικότερη ε, εικόνα, να δούμε δηλαδή στις λεπτομέρειες ποια προληπτικά μέτρα απαιτούνται, π.χ. Ναι, η εργασία με τα ρομπότ που δεν είναι πλέον ε, εγκλωβισμένα. Τι σημαίνει αυτό για την υγιεινή και την ασφάλεια. Εργασία με τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο είναι το αφεντικό, ποιο λαμβάνει τι αποφάσει. Υπάρχουν διάφορε πτυχέ ε, λοιπόν και αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσουμε μετά την οριστικοποίηση αυτή της ε, πτυχής αυτού του έργου για μια εκστρατεία ε, γίνεις στο χώρο εκστρατείας. Η επόμενη σχετική εκστρατεία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τις μειοσκελετικές ε, παθήσεις, ε, το οποίο το σχετίζουμε με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και υπάρχει ένας κίνδυνος πάρα πολύ σημαντικός. Βλέπουμε όλο και περισσότερες ασθένειες ψυχικές που σχετίζονται με την εργασία. Μειοσκελετικές ασθένειες λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικές, είναι μια αιτία για μακροχρόνια άδεια και για πρόορη συνταξιοδότηση και ήδη έχουμε προετοιμάσει ένα μεγάλο έργο που αφορά διάφορες πτυχές ε, των μειοσχηλετικών ασθενειών και του χρόνου θα ξεκινήσουμε μια καμπάνια για την υγιεινή στο χώρο εργασίας που αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Επίση, ε, αυτό το οποίο ανέφερε και η κυρία Φαντεμπέλεν είναι ένα οριζόντιο θέμα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το πώς θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εταιρείες και βέβαια η πτυχή του φύλου. Μετά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο ανέφερε ένας συνάδελφος, δηλαδή το πώς έχουν τα πράγματα με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας. Το ανέφερα και πριν, είμαστε μοναδικοί, δηλαδή είμαστε ένα δίκτυο εμείς, δηλαδή είμαστε σε συνεχή επαφή με τα 28 κράτη-μέλη, μόλις επέστρεψα από τη Σλοβενία την προηγούμενη εβδομάδα, και εκεί πέρα ακριβώς έχουμε την ενημέρωση από το δίκτυο αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά όπως ανέφερε και ο Χάν και οι συνάδελφοί ε, έχουμε και έρευνες που γίνονται τακτικά και βεβαίως να αναφέρω εδώ πως ε, το αποτέλεσμα αυτό ήταν πολύ θετικό πάνω από 90% των ενδιαφερμένων και των συμμετεχόντων να χρησιμοποιούν το υλικό μας, τις δραστηριότητές μας στην καθημερινή τους ζωή, στην εργασία τους. Και τέλος, α, βεβαίως, αυτό το οποίο ανέφερα, ναι, βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ψυχικές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και θα ήθελα να πω πως Τώρα οι μελλοντικέ μας προβλέψεις ε, αφορούν ακριβώς και τον αντίκτυπο ε, στην υγεία, τον ε, ψυχοκοινωνικό κίνδυνο και τώρα βεβαίως θα έχουμε και την εργασία στο διαδίκτυο με την τεχνητή νοημοσύνη οπότε θα δούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω τι σημαίνει αυτό για την υγεία. Τελευταίο σχόλιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης μας για τους νέους κινδύνους και φέτος ρωτάμε εταιρείες ε, όλων των μεγεθών και φέτος περιλάβουμε για πρώτη φορά και τις, ψυχε, τις πτυχές της ψηφιοποίησης. Δηλαδή για πρώτη φορά θα δούμε ποια είναι η αποδοχή της, πώς χρησιμοποιείται και ποιες είναι οι προκλήσεις και νομίζω μέχρι το τέλος του έτους θα γνωρίζουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ο κύριος Ωνεστίνη θα κλείσει τον πρώτο κύκλο απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα που νομίζω έχουν σημασία για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης. Πρώτα απ' όλα για τον κοινωνικό πυλώνα. Ακόμα και να εργαζόμαστε με τρίτες χώρες, το γεγονός ότι η πρώτη αρχή του πυλώνα αυτού είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση και διαβίου κατάρτιση μας δίνει μια ισχυρή εντολή και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Αναφέρθηκε η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ε, στην εκπαίδευση, αυτή είναι η πρόκληση ε, ο σύνθημα βεβαίως υπάρχει εδώ και καιρό ως πολιτική νομίζω είναι κάτι το οποίο ακόμα αναζητούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αλλά στις ε, χώρες ε, τερούς ειδικά στη γειτονιά που δουλεύουμε βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις προσεγγίσεις και το πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε διάφορα παραδείγματα του πώς εργαζόμαστε και ακριβώς έρχομαι στο πόσο ικανοποιημένοι είμαστε. Εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά εάν από την ε, πλευρά μας καταφέρουμε να έχουμε στοιχεία και να έχουμε περισσότερα στοιχεία για να έχουμε ακριβώ μια τέτοια προσέγγιση σε ένα περίπλοκο τομέα πολιτικής αλλά και το πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που λαμβάνουμε ε, με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα στον διάλογο με τις ε, χώρες και δεύτερον σε προγράμματα και έργα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι σε όλες τις χώρες του δουλεύουμε ο μεγαλύτερος πάροχος ε, στήριξης ε, και νομίζω ότι και στις δύο πτυχές σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο ειδικά όσον αφορά τον διάλογο πολιτικής με τη Γενική Διευθύνση Απασχόλησης έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε πολύ στενότερη επαφή μεταξύ των όσων παρέχουμε στα κράτη-μέλη και το πώς ε, τα κράτη-μέλη εξάγουν τον διάλογο πολιτικής. Οπότε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε κάποια καλά παραδείγματα του πώς ε, η δουλειά που κάνουμε στις χώρες μετά χρησιμοποιείται στο πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο των έργων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε υπάρχουν αρκετά ονόματα ομιλητών. να σε ρωτήσω αν μπορούμε να ορίσουμε τον χρόνο ομιλίας στα δύο λεπτά. Ανά ερώτηση. Να πω τα ονόματα. Madam Sparentak, Madam Sparentak, Madam Zalewska, Madam Zdanoka, Mr. Patton, Mr. Forles, uh, Mr. Kanev, Mr. Lenars,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 για τι πολύ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει. Έμαθα πολλά ω νέο ευρωβουλευτή. Έχω όμως μια συγκεκριμένη ερώτηση για την κυρία Σέντλατσεκ όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας. Πρώτα απ' όλα, πώς θεωρείτε ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη δράση και συνεργασία μεταξύ των ε, κρατών μελών και πώς ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Συγκεκριμένα για τις επικίνδυνες ουσίες ε, στο χώρο εργασίας έχουμε τον γνωστό κανονισμό REACH ε, για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που θα έπρεπε να δούμε τα μείγματα επίσης που υπάρχουν στην αγορά και βεβαίως δεν ε, χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση μετά την αγορά γιατί έχουμε ήδη την αξιολόγηση πρώτης αγοράς αλλά όπως έχουμε για τα φάρμακα ή τις ιατρικές συσκευές ή άλλα καταναλωτικά προϊόντα δεν χρειάζεται και εδώ μια τέτοια εποπτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σπάρντακ, η δική σας ερώτηση και η κυρία Ζαλεύσκα να ετοιμάζεται. Σας ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Η πρώτη απευθύνεται στην Σεντεφόπ. Ε, το πράσινο New Deal βεβαίως ε, θα είναι σημαντικό για την ε, δουλειά της Κομισιόν και ελπίζουμε να φέρει ευημερία για όλους. Γι' αυτό είμαι για το εάν προετοιμάζετε κάποια εργαλεία για να προβλέψετε την πράσινη μετάβαση και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν για το Eurofund. Με χαρά είδα την δημοσίευση της έκθεσης για την εργασία στις πλατφόρμες, όπως είπατε, και λέει εκεί ότι ε, μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε εργασία χωρίς ε, εμπόδια και μπορούν εκεί πέρα να απασχοληθούν ευάλωτες ομάδες. Αλλά ε, ακριβώς γι' αυτό είναι ενισχυτικό το ότι ένα άλλο έβριμα ήταν ότι κανένα κράτος μέλος δεν έχει σαφείς κανόνες για το καθεστώ απασχόληση των εργαζομένων αυτών. Ε, κάτι το οποίο είναι ίσως ε, κίνδυνο για τα εργασιακά δικαιώματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν να θα συνεχίσετε να εργάζεστε επί του θέματος και ε, ίσω αν κάνετε κάποιε συγκριτικέ μελέτες για το πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό για να δούμε και πώς μπορεί να ξεκαθαρίσει το καθεστώς τους και προς την όσα επίσης πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα προστατεύονται από την σκοπιά της ασφαλείας και της υγιεινής. Σας ευχαριστώ η κυρία Ζάλευσκα και ετοιμάζεται η κυρία Σντάνοκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το ότι συνεδριάζουμε και μιλάμε για το μέλλον ε, των υπηρεσιών αυτών οφείλεται ακριβώ στην δουλειά της Προέδρου. Έχουμε τις προκλήσεις που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια βεβαίω. οπότε έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα, όταν εσείς κυρίες και κύριοι παρουσιάζετε την δουλειά σας και έχουν εντύπωση ότι εργάζεστε παράλληλα και όχι μαζί για να κάνετε κάποιες κοινέ εκθέσεις Επίσης ε, δεν βλέπω να μιλάτε για τον αντίκτυπο, τα αποτελέσματα που έχουν οι εκθέσεις σας. Η διεξαγωγή των μελετών, ε, ε, οι, οι αναφορές, οι παραπομπές. εντάξει νομοθεσία ε, εδώ πέρα και οι εκθέσεις εδώ πέρα πράγματι θα επηρεάσουν τον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς. Ε, ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και τα αποτελέσματα συχνά είναι άσχημα και είναι δύσκολο να συγκρίνουμε διάφορες ε, χώρες. Προφανώς γνωρίζω καλύτερα την Πολωνία. Στην Πολωνία η κατάρτιση είναι κακής ποιότητας, είναι λίγα τα μαθήματα, μακριά από τους εργαζόμενους, είναι για ενηλίκους που είναι ήδη εκτός του συστήματος. Ή τρέπονται που δεν έχουν δεξιότητες ε, κτλ. Οπότε πώς ε, μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο για να αλλάξει αυτό. Το ένα είναι αυτό. Μετά, για την εξατομίκευση. Ε, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε τα ονόματα των ερευνητών που κανάζει. Αυτά και θα κάνω όλες τις ερωτήσεις μετά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σντάνοκα και να ετοιμάσω κύριο Σπάτσον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Έχω ερώτηση και ένα σχόλιο προς τον κύριο Μενέντες Βάλτες. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα ευρήματά σας, τα χρησιμοποιήσαμε στην έκθεση για την ε, ισορροπία ζωής ε, και εργασίας, ε, στην οποία ήμουν εισηγητρία. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για τον βασικό μισθό αναφέρθηκε. Είχαμε διάφορες προτάσεις. Γνωρίζω πως έχετε πρόσφατα ευρήματα θα κάνετε κάποιες συστάσεις επίσης για, και για το ελάχιστο εισόδημα, όχι μόνο το βασικό μισθό και ένα άλλο θέμα η στέγαση. Η έρευνά σας ε, το κοιτάει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και ο Σαπάτεν και ο κ. Φούρλας να ετοιμάζετε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις έχω η πρώτη αφορά την επαγγελματική κατάρτιση μου προξένησε. εντύπωση ε, πολλά σχόλια. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και συχνά το υποτιμούμε. Ε, ποια δουλειά έχετε κάνει λοιπόν, όχι μόνο με κράτη και κυβερνήσει, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών και μικρές ε, οργανώσεις που είναι σημαντικές και καλύτερες θα έλεγα από ε, μεγάλα θεσμικά οργανά στον φτάνουν σε ε, ομάδες που δύσκολα μπορούν να φτάσουν άλλοι. Το άλλο μου ερώτημα αφορά το ETF. Μήπω ε, τη δουλειά σας θα την έκανα καλύτερα τα κράτη-μέλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα διεθνή οργανισμός όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι τέτοιο. Η τρίτη μου ερώτηση είναι πιο προσωπική. Ε, και να με συγχωρείτε, έχω αρχίσει να βαριέμαι να κοιτάω πάνελ ε, σχεδόν αποκλειστικά έτσι, τέτοιας ε, σύνθεσης. Ε, εντάξει, επικροτώ την δουλειά που γίνεται όσον αφορά το φύλλο, αλλά τι κάνετε όσον αφορά τις φιλετικές μειονότητες, όσον αφορά την έρευνα που υπάρχουν ουσιαστικές ανισότητες και έλλειψη εκπροσώψης. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξουν κάποια σχέδια ως προς αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποφεύγει. Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Όταν προσέθεσα τα νούμερα, ε, βρήκα συγκεντρωτικά ότι εκπροσωπείται ε, ε ουσιαστικά έναν προπολογισμό 125 εκατομμυρίων ευρώ. Κάποιοι ρωτήσαμε το τι αντίκτυπο έχετε και έχετε δώσει κάποιες ε, σωστές απαντήσεις όσον αφορά την έρευνα και τις παραπομπές, αλλά αισθάνομαι και κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι ε, δεν είναι σωστή λογοδοσία αυτή σε σχέση με τους στόχους που έχετε. Το ερώτημά μου είναι τα 125 εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύουμε για σας ε, θεωρείτε ότι έχουν διατεθεί σωστά. Ο κύριος Φούρλας και ο κύριος Κάνιεφ να ετοιμάζεται. Διότι σήμερα εμείς οι νέοι ευρωβουλευτές μάθαμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σταθώ στο σημαντικότερο νούμερο που έχω ακούσει σήμερα. Και η ερώτηση μου απευθύνεται στην διευθύντρια ε, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Ευρώπη, 150.000 άνθρωποι νεκροί κάθε χρόνο στην Ευρώπη από ασθένειε που σχετίζονται με την απασχόληση. Φωνιά ο καρκίνο, έχετε πει. Και το ερώτημα μου είναι κατά πόσο θα συνεργαστείτε μαζί με την νέα πρόεδρο τη Κομισιόν, η οποία θέλει να ελοποιήσει το πρόγραμμα για την καταπολέμηση του καρκίνου σε πενταετέ ε, πρόγραμμα ε, έχω ακούσει επίσης ότι έχετε ένα εργαλείο το οποίο αξιολογεί την επικίνδυνοτητα, το οποίο είναι και δωρεάν, κατά πόσο αυτό χρησιμοποιείται από τον κόσμο, δηλαδή σε ποιο βαθμό υπάρχει πρόσβαση ε, και χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Και μεταφέρω και ένα ερώτημα από τον συνάδελφο τον Στέγιο τον Κιμπουρόπουλο, ο οποίος έπρεπε να φύγει. Πώς μετράτε το εργασιακό burnout και αν βλέπετε παρατυπίες, αν έχετε δυνατότητα να επιβάλλετε κάποιες κυρώσεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Κύριος Κάνιεφ και ο κύριος Λενάρχς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Για τη ΣΕΝΤΕΦΟΠ είναι η ερώτηση περισσότερο. Συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που καταβάλλετε για την επαγγελματική κατάρτιση και τις προσπάθειες για καλύτερα, καλύτερη πρικοδότηση για την επαγγελματική Σε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία όμω ε, υπάρχει αύξηση των ανισορροπιών. Η αγορά εργασία πεινάει για προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και πιο ευάλωτες ομάδες, κυρίως η μειονότητα των Ρωμά, μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Είτε λόγω μόνιμης ανεργίας, είτε λόγω εργασίας στην κρίζα ζώνη, είτε στη Βουλγαρία, είτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ολόκληρες περιοχές και χώρες ταυτόχρονα είναι οικονομικά ανταγωνιστικές μόνο λόγω χαμηλών αμοιβών που παρέχουν. Δύο ρωτήσεις. Η πρώτη. Λόγω διοικητικής και οικονομικής προσπάθειας θα έπρεπε να καταβληθεί παράλληλα και νομοθετική προσπάθεια, όντως ώστε η επαγγελματική κατάρτιση και η απασχόληση να διασυνδεθούν καλύτερα σε όλη την Ευρώπη. Άλλη ερώτηση. Πώς αξιολογείτε τη σχέση μεταξύ ελάχιστου εισοδήματος ή ελάχιστης εισφοράς για τις ασφάλειες και αγορά εργασίας για τις ευάλωτες ομάδες. Ο κύριος Λέναρς και η κυρία Φερνάντες μετά. Ευχαριστώ. Λέει ο κ. Εδώ και ένα μισή χρόνο, Επίτροπο Τάισαν παρουσίασε την πρόταση για την ΕΛΑ. Χαίρομαι που μετά από 1,5 χρόνο, μόλις μετά από 1,5 χρόνο, έχουμε το διευθυντή της ΕΛΑ για να παρουσιάσει τις δραστηριότητε του οργανισμού. Τεράστιο πίτευμα που πιστώνεται στην Επίτροπο Τάισον και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ρουμανική Προεδρία και πολλούς συναδέλφους, συμβούλους και βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάστηκαν σκληρά ούτω ώστε να καταστήσουν εφικτό. Και έχουμε ευθύνη σαν Κοινοβούλιο να διορίσουμε εμπειρογνώμονα που θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα έχει φωνή. Με τα χαράς βλέπω επίσης και την πρώτη δημοσίευση έξι κενών θέσεων από 2004 και ζήτησαν να είναι υποψήφιοι 2.400 άνθρωποι για να εργαστούν στον οργανισμό. Ελπίζουμε να είναι εξίσου δημοφιλής για τις προσλήψεις όσο και για τις δράσεις που θα δρομολογήσει. Είναι μοναδική ευκαιρία που έχουμε εδώ όλους τους φορείς μαζί. Ο κανονισμός για το ΕΛΑ είναι σαφής. Πρέπει να έχει στενή συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς για κοινωνικά θέματα και απασχόληση. Να δημιουργηθούν συνεργασίες και να αποφευθούν επαναλήψεις και αλληλεπικαλήψεις. Τι συγκεκριμένα σχέδια υπάρχουν στους άλλους οργανισμούς και στον ΕΛΑ, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό. Το έργο του ΕΛΑ να είναι προστιθέμενη αξία στις εργασίες των άλλων ε, φορέων και πώς υπάρχει συνεργασία στο μέλλον. Κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις Νομίζω ότι εμφεθήκαμε σε θέματα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων. Να αναφερθώ σε κάτι που συζητήθηκε. Θέλω να υπογραμμιστεί. Συνθήκες εργασίας και κυρίως η υγεία στα πλαίσια του τόπου εργασίας. Στην, ε, στην Επιτροπή Απασχόληση ε, προβληματιζόμαστε. διότι τα κοινωνικά θέματα έχουν μοιραστεί σε διάφορα χαρτοφυλάκια η απασχόληση δεν έχει ενταχθεί στο ίδιο με τα κοινωνικά θέματα. Προσπαθούμε να πετύχουμε επιτεύγματα σε διάφορα θέματα όπως είναι η υγεία στον τόπο εργασίας. Όλοι εδώ οι οργανισμοί που είναι παρόντες και εκπροσωπούνται, κυρίως το Eurofound, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Εμείς οι σοσιαλιστές ε, ζητήσαμε ο Νίκολας Μιφ, από τον Νίκολα Σμιφ ζητήσαμε να επιμείνει επί του γεγονότος να μην αναφέρονται στο χαρτοφυλάκιο του κοινωνικά θέματα. Του ζητήθηκε αυτό. Θα ήθελα να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών Eurofound και οσά με τον αρμόδιο πίτροπο που θα είναι υπεύθυνο για απασχόληση για θέματα που είναι σημαντικά εργάζεστε πολύ για τα θέματα της υγείας, το ξέρω. Και πρέπει να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. Και το Eurofound είναι στη βάση της έννοιας της βιώσιμης απασχόλησης. Χρειάζεται πολυδιάστατη προσέγγιση, όπως είπε και ο Μενέντες Βάλτες. Μόνο με πολυσχηδή προσέγγιση μπορούμε να οδηγηθούμε σε βιώσιμη ανάπτυξη να έχουμε βιώσει με στέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ και βασίζομαι στη συνεργασία κυρία Μπρουνέν, ετοιμαστή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις και δόθηκαν και αρκετές απαντήσεις. Αυτά συμβαίνει όταν κανείς μιλάει τελευταίο στο δικό μου το ερώτημα πηγαίνει προς την κατεύθυνση των ασθενειών της πλάτης αναφερθήκατε κυρία στα μειοσκελετικά μπορείτε να αναφερθείτε στην πρόληψη το παράγοντα του κόστους και αναφέρατε επίσης ότι Υπάρχουν κάποιες μελέτες, ε, κατάλαβα καλά, και έργα τα οποία ε, θέλετε να υλοποιήσετε. Αν δεν έχω καταλάβει καλά, διορθώστε με. Γιατί ήταν πολύ συναρπαστικό αυτό το οποίο είπατε. Ποια είναι συγκεκριμένα όμως τα σχέδια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε εδώ πέρα την κατάσταση ε, πιο ενεργά γιατί όπως είπαμε οι θέσεις εργασίας ε, δημιουργούν πραγματικά ένα θέμα όσον αφορά ακριβώς τους ε, τραυματισμούς στην πλάτη. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Μπρούνε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Μία ερώτηση έχω. με τον κύριο Μενέντε Βάλτας, τον κύριο Σίπελ και τον κύριο Ονεστίνη. Πρόσβαση στην κατάρτιση, κυρίως από πλευράς γυναικών. Είναι ένα θέμα που έχουμε στη Γαλλία, όπου οι γυναίκες μπαίνουν λιγότερο στην επαγγελματική κατάρτιση τη διάρκεια της ζωής. Είναι ένα από τα αίτια των μισθολογικών διαφορών στην επαγγελματική ζωή. Θα ήθελα απάντηση επ' αυτού του συγκεκριμένου. Δεύτερη ερώτηση. Εν μέρει ετέθη προς την κυρία Σελατσέκ. Τις μελέτες που κάνατε για τον κίνδυνο για την υγεία, κυρίως τους εργαζόμενους της πλατφόρμας. Για τα προβλήματα δηλαδή που εντάσσεται στα προβλήματα της υγείας στον τόπο εργασίας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στους φιλοξενούμενούς μας. Η κυρία Σέντλατσεκ. Καταρχάς, οι περισσότερε ερωτήσει αφορούσαν εσά και την όσα. Και μετά θα πάμε στον κύριο Βάλτε. Η κυρία Σέντλατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει σας. Πολύ ενδιαφέρουσε, Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας την πρώτη ερώτηση που αφορά στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η άποψή μου είναι αυτή και η εμπειρία του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτή, αν δεν έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία στον τόπο απασχόλησης, το εθνικό επίπεδο θα αναμένει αυτή τη στρατηγική. Και ξεκινούν οι κοινωνικοί, τις επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο κρατών να δουν την τελική εκδοχή στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα στατηγική της ευρωπαϊκή Ενώσεως εκπνέει το 2020. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη άρχισαν συζητήσεις. Μπορώ να πω ότι σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται ένας προσανατολισμός. Οι βασικές προτεραιότητες για την ασφάλεια στον τόπο εργασία που θα συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του κοινωνικού εταίρου. Η εμπειρία που είχαμε ποια ήταν. Ότι μετά ακολουθούν και βλέποντας τις τρέχουσες στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο, λίγο πολύ όλες αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θετικό να δοθεί συνέχεια στη στρατηγική. Επικίνδυνα χημικά. Περίπλοκο ερώτημα. Αναφερθήκατε στον κανονισμό το σχετικό με το REACH, την εκ των προτέρων αξιολόγηση εντός των σχετικών κανόνων και οι περισσότερες διατάξεις αφορούν ουσίες και όχι μείγματα. Αυτή δεν είναι η περιοχή πολιτικής μας. Δεν ασχολούμεθα με αυτή την νομοθεσία. Συνεργαζόμαστε όμως με την ΕΚΑ. Προσωπική άποψη εκφράζω. Διότι η άποψη αυτή οδηγεί και στον τόπο εργασίας. Και εκεί είναι παρόμοια η κατάσταση. Εκείνοι που παράγουν ένα προϊόν πρέπει να ενημερώνουν τον εργοδότη για όλα τα συστατικά και την τελική χρήση. Ο εργοδότης υπέχει υποχρέωση επίσης να ενημερώσει τον παραγό του προϊόντος για άλλες χρήσεις, άλλες περιστάσεις ή υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν λειτουργεί όμως στην πράξη. Εμείς, όσον αφορά τόπο εργασίας, πρέπει να εξετάσουμε την ύπαρξη ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων που αφορά τη χρήση και τον αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων. Είχαμε ένα δημοσίευμα για ένα σύστημα επιφυλακής και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν αυτά τα συστήματα σε εθνικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ένα φερρυπίν. Χρησιμοποιείται ένα προϊόν σε μια εταιρεία. Και ας πούμε προκαλεί αλλεργία. Ο οικογενειακός γιατρός το ανακαλύπτει πρώτος. Ή ο γιατρός, ο γειτονικός σε πανεπιστήμια σχεδόν σε όλες τις χώρες από ό,τι ξέρουμε οι γιατροί δεν έχουν εκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση υποχρεωτική για την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας. Οπότε οι αναφορές αυτές καταλήγουν οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει απόδειξη συγκεκριμένη για την αλλεργία που συνδέεται με συγκεκριμένο προϊόν είναι λογική η, μετά την χρήση να, αξιολόγηση να γίνεται, όπως μετά τη διάστηση αγορά. Άρα πρέπει να γίνει ανάλυση του θέματος και πολλή κουβέντα. Και άλλες ερωτήσεις για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Είχαμε κάποιες αστηριότητες προετοιμασίας και για την ψηφιοποίηση Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στην ιστοσελίδα μας. Τι είναι το πιο σημαντικό. Όλοι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους λίγο πολύ, όπως μια καθαρίστρια που εκτίθεται σε μια εταιρεία ή σε μια οικοδομή. Σχεδόν το ίδιο, αλλά οι περιστάσεις και η πρόσβαση στους εργαζομένους αυτούς είναι πιο δυσχερής. Άρα χάνουν, μη λείπει ο έλεγχος, η πρόσβαση στις υπηρεσίες όσα και στα προληπτικά μέτρα. Εκεί είχαμε ετοιμάσει στις Βρυξέλλες πέρσι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο. Προσεκλήθησαν πολλοί εμπειρογνώμονες από πολλά κράτη-μέλη και παρουσίασαν την προσέγγιση τους. Δηλαδή, πώς να υπάρξει η πρόσβαση ή να ρυθμιστεί η εργασία στις πλατφόρμες, μπορώ να σας παραπέμψω σε αυτά τα αποτελέσματα, διότι όλες οι χώρες έχουν διαφορετική προσέγγιση. Η Γαλλία έχει προχωρήσει περισσότερο. Το Ηνωμένο Βασίλειο κάτι κάνει, αλλά ανάλογα με τα συστήματά τους και τις ανάγκες τους. Και δεν υπάρχει μια γενική λύση αλλά σύμφωνα με τι ανάγκε. Είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανεί προσεγγίσει των διαφορών χωρών. Ποιο είναι το σημαντικό όμω, να συνεχιστεί η συζήτηση με τα κράτη-μέλη, κυρίω η συζήτηση με του κοινωνικού εταίρου, διότι έχουν τη δική του στρατηγική. Να βρεθεί μια τελική λύση. Μέτρα συμπεφωνημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες. Πηγαίνετε στο σελίδα μας παρακαλώ να δείτε τις μελέτες και τη συνέχεια που δίδεται στα απορίσματα. Κάτι άλλο αναφέρθηκε. Κάποιο σχόλιο ακούστηκε. Αν συνεργαζόμαστε, είπατε δεν συνεργαζόμαστε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν εργαζόμαστε έτσι. Συμφωνούμε κάθε χρόνο. Και προσυπογράφουμε ένα υπόμνημα για τη συνεργασία μας σε ποιους τομείς θα συνεργαστούμε για να αποφευχθεί η αδίποτε επικάλυψη. Καλά τα πάμε. Είναι περίπλοκο το θέμα υπιοποίησης. Είναι μια ανάγκη. Έχουμε ασφάλεια και γίνει στον τόπο εργασίας και εδώ μιλάμε για όλο τον κοινωνικό τομέα. Χρησιμοποιούμε όμως όλες τις μελέτες. Αν δείτε τις μελέτες μας και του Eurofound, θα δείτε ότι χρησιμοποιούμε τις μελέτες μας το πρώτο που κάνουμε είναι εξετάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Ε, είμαι ανοιχτή όμως. Μπορώ να αναφέρω λεπτομέρειες. Ίσως να μην διαβιβάζουμε με επαρκή τρόπο τις πληροφορίες. Το ερώτημα, το θέμα του καρκίνου που θέσατε, ναι, είναι μια καταστροφή, αν δείτε τους αριθμούς, καταστροφικά αποτελέσματα. Υπέχουμε υποχρέωση ηθική να προλάβουμε την εμφάνιση του προβλημάτος. Και πρέπει να δούμε και το κόστος όλων των ασθενειών και των θανάτων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όσον αφορά τον καρκίνο, να συμμετέχουν πολλοί κοινωνικοί εταίροι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάφοροι οργανισμοί και υπηρεσίε. Η Φιλανδία και τα άλλα μέλη συμμετέχουν. Μια σημαντική πρωτοβουλία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της Ολλανδίας έλαβε χώρα. Ξεκίνησε η καταπολέμηση του καρκίνου. Μια μεγάλη πρωτοβουλία δρομολογήθηκε. Και τώρα όλες οι προεδρίες, όπως η Φινλανδική Προεδρία, μετά η Γερμανική Προεδρία, θα ηγηθούν της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση του καρκίνου. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, συνεργασία, έρευνα που γίνεται στον τομέα και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει το πώς θεωρείται σημαντική η καταπολέμηση του καρκίνου. Πάρα πολύ σημαντική. Αναφερθήκατε την αξιολόγηση, το εργαλείο ή την αξιολόγηση του κινδύνου στο διαδίκτυο. Ναι, είναι ένα εργαλείο όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, χωρίς κανένα κόστος, δωρεάν, για πολλούς τομείς, για πολλά καθήκοντα είναι πραγματικά εύκολος κατάλογος, μια λίστα που μπορεί να τη δει ο καθένας και θα ήθελα ίσως, γιατί πρέπει να σας εξηγήσω λίγο πώς να έχετε πρόσβαση, διότι υπάρχουν σημεία επαφής, αλλά δωρεάν διατίθεται. Για το burnout και την ασυνήθιη εργασία Μέχρι το έτος 2008 κάναμε έρευνες, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλες έρευνες έγιναν και έδειχαν τον ψυχοκοινωνικό κίνδυνο που αυξάνονται αυτοί οι κίνδυνοι. Αναφέρθηκε και αυτή η υπερκόπωση, το burnout, που αναφέρεται στις έρευνες μετά το 2008 και τα επόμενα έτη. Τι άλλο. Έμεστη, η κυρία Φερνάντες. Θέλατε κάποια απάντηση ή είπατε ότι πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι, ήταν σχόλιο περισσότερο. Όχι, όχι, λέει και Φερνάντες. Όχι απάντηση. Χρειάζεται όμως να, ε, οπωσδήποτε να συνεργαστεί το Κοινοβούλιο με αυτές τις δικές σας ε, οργανισμούς ώστε να καλύψουμε τα πολύ σημαντικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, αυτή η, ο πόνος στην πλάτη, τα προβλήματα τα ραχεία, τα προβλήματα της πλάτης, ξεκινήσαμε να εξετάζουμε τα μειοσκελετικά προβλήματα, τους διάφορες παράγοντες, διάφορες παράγοντες που, που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα τα μυοσκελετικά, τον πόνο στην πλάτη. Κάθε δεύτερο ένα στους δύο στην Ευρώπη έχει προβλήματα με την πλάτη του κατά τη διάρκεια της ζωής του. και σε αυτό το πρόγραμμα για τους μειοσκελετικούς κινδύνους και τα προβλήματα. Δίνουμε ένα συγκεκριμένο, τονίζουμε ιδιαίτερα τα προβλήματα της πλάτης, τον πόνο της πλάτης και πώς μπορεί να επιστρέψει κανείς την εργασία του. Πολλοί παίρνουν μακροπρόθεσμες άδειες λόγω μειοσκελετικών προβλημάτων, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση πριν φύγουν με άδεια και μετά πώς να επιστρέψουν την εργασία τους και πώς να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν ξανά. Και άλλες τυχές ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Ξέρουμε ότι εκείνοι που εργάζονται σε χώρους με ένταση, με στρες, αναπτύσσουμε σκελετικά προβλήματα, κυρίως πόνο στην πλάτη. Θα δείτε τα αποτελέσματα υπάρχουν, αλλά και συστάσεις για επιχειρήσεις, για εργαζομένους, για εκεί που την πολιτική να βελτιώσουν την κατάσταση. Και τώρα ξεκινά μια εκστρατεία για μυοσκελετικά προβλήματα του χρόνου θα ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για όλο το θέμα και θα συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο επίσης να διαδοθεί το μήνυμα, να περάσει το μήνυμα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει λίγο τον χρόνο και χαίρομαι που είστε τόσο ε, ενεργός. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω και άλλη ερώτηση όμως. Δεν ήθελα άλλη ερώτηση. Ε, να πω μόνο ότι έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Ε, σέβομαι τους ομιλητές, αλλά έχουμε και σημαντικά θέματα μετά. Και θέλω να μιλήσω και στο επόμενο. Ναι, ναι, μην ανησυχείτε. Αυτό ακριβώς ε, αυτό θα έκανα, κύριε Πάτεν. Α, πρέπει να βάζω και κάποια χρονικά ώρα για τις απαντήσεις, γιατί είναι άδικο βεβαίως. Δεν είχα βάλει χρονικό όριο να σας παρακαλώ να είστε ως το δυνατόν πιο σύντομοι και όποιος ε, και δώσει τη συντομότερη απάντηση κερδίζει χρυσών ορολόγιων. Λοιπόν, ε, ο κύριος Βαλντέζη και να ετοιμάζεται ο κύριος Ανεστίνη. Ωραία, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε μια ερώτηση για τα ζητήματα συνεργειών και λογοδοσίας προς το Κοινοβούλιο. Μια σωστή ερώτηση γιατί βεβαίως πρέπει να λογοδοτούμε. Έχουμε λοιπόν αυτή την συνεννόηση με τις άλλες υπηρεσίες, ανταλλάσσουμε τα προγράμματα πριν εγκριθούν, συμφωνούμε με κοινέ δραστηριότητες, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ερευνατών Εταιριών, έχουμε κοινέ εκθέσεις για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που ανέφερε η κυρία Φερνάντες και έχουμε και άλλα στοιχεία. Αντίκτυπο. Ναι, έχουμε αντίκτυπο στην ομοθεσία, όχι άμεσο, γιατί ε, δεν είμαστε πολιτικοί φορείς, εμείς σας δίνουμε τα στοιχεία εσείς είστε οι πολιτικοί, μπορείτε όμως να δείτε την χρήση των ευρημάτων μας στην οδηγία για την ισορροπία εργασίας και ζωή, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, στην εγγύηση για την νεολαία, βεβαίως το πόσα λεφτά. Ε, λογικό να το λέτε. Νομίζω ότι ε, τα τελευταία χρόνια περάσαμε μία μείωση του προσωπικού κατά 10%. Βλέπουμε ε, κυβερνήσεις να ζητάνε όλο και περισσότερα πράγματα από εμά γιατί χρειάζονται συγκριτικές ε, πληροφορίες ε, που δεν έχουν γιατί έχουν τις εθνικές και είναι κρίμα το ότι βλέπουμε κάποια πράγματα παραδείγματο χάρη είναι κρίμα το ότι βλέπουμε τη σύγκριση του Ηνωμένου Βασιλείου με άλλες χώρες Είμαστε υπόλογοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι κυβερνήσεις σας υπολογιστήν ε, κομισιόν επίσης ε, ε, υφιστάμεθα διαφόρους δημοσιονομικούς ελέγχους και ερχόμαστε για την απαλλαγή στο Κοινοβούλιο που νομίζω ότι για το μέγεθος του οργανισμού μας ο έλεγχος που υφιστάμεθα είναι πολύ μεγαλύτερος από ένα δήμο ξέρω που έχει ανάλογο μέγεθος. για τα θέματα των πλατφορμών, σωστά είπατε, έχουν θετικές και αρνητικές πτυχές. Είναι διαφορετική η κατάσταση, κάποιες είναι κάπως πιο ύποπτες, άλλες έχουν σαφώς μια ξεκαθαρή λειτουργία. Έχουμε επίσης συνθέσει όλη την έρευνά μας, όχι μόνο για εμάς στην ιστοσελίδα μας, οπότε δεν θα τα αναπτύξω τώρα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, όχι μόνο κανονισμός, ε, συλλογικές συμβάσεις και εθελοντικά μέτρα, μεταξύ άλλων, για το θέμα του βασικού μισθού και τις ε, συστάσεις ε, τηλεγραφικά πρέπει να δούμε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση σε κάθε χώρα, εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, Απολύτω απαραίτητο όταν μιλάμε για καθορισμό μισθών και βεβαίω ένα διαφανέ ε, σύστημα. Έχουμε 22 χώρε που έχουν βασικό μισθό, δύο που το συζητάνε. Έχουν χώρες που δεν θέλουν να έχουν κάτι τέτοιο γιατί έχουν άλλες ε, λύσεις, ε, δηλαδή συλλογικέ συμβάσεις όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες ή η Αυστρία. Το θέμα της ισορροπίας ζωής και εργασίας το αναφέραμε ήδη. Είπα κάτι πριν, οπότε σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Ωνεστίνη και να ετοιμάζεται ο κύριος Ζίπελ. Ε, ευχαριστώ. Τρία σύντομα σημεία. Ε, ένα για το θέμα της συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε στενά με το Σεντεφόπ και το Eurofound για λόγους μεθοδολογίας και τα λοιπά. Ε, μετά αποκλίνουμε στον τρόπο εφαρμογής, οπότε υπάρχει κάποιο όριο στο τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Δεδομένου του ότι η εντολή είναι διαφορετική στην περίπτωσή μας να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπατε για το φύλλο και τα σχετικά το οποίο το βλέπουμε στις χώρες μας η συγκριτική πτυχή είναι ενδιαφέρουσα γιατί βλέπουμε ότι παρά το ότι κάποιες χώρες κάνουν κάτι το ζήτημα υπάρχει ε, οπότε νομίζω ότι η απάντηση πηγαίνει βαθύτερα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα που προσπαθούμε να δούμε και να δούμε αυτή την διάσταση της επιλογής όταν είναι επιλογή ε, του φίλου για να μπει στην προσπάθεια της μεταρρύθμισης και τέλος το θέμα του σκεπτικού των δράσεων αυτών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης ε, ε, έχει φτιαχτεί για να στηρίξει την ευρωπαϊκή εξωτερική δράση που θεωρείται ότι επηρεάζει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες τις άλλες. Ε, δεν υποκαθιστά τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη και θέλω να τονίσω μάλιστα ότι σε κάποιες από τις χώρες που εργαζόμαστε τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ ενεργά. Έχουμε πολύ ε, στενή συνεργασία μαζί τους ε, και βεβαίω είναι γνωστό ότι υπάρχουν συνέργειες αλλά είναι αλήθεια ότι δεν δραστηριοποιούμαστε σε όλες τις χώρες και υπάρχει μια συστημική προσέγγιση στα όσα κάνουμε τελικά ε, θέλουμε να έχουμε μια πιο σταθερή γειτονιά, γιατί να μπορούν οι χώρες αυτές να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να στηρίζουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κοινό ε, καλό και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Εκεί πέρα συνεισφέρουμε. Σας ευχαριστώ. κύριο Ζίμπελ ε, και ο κύριος Κορέλ να ετοιμάζεται. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα εστιάσω το πράσινο New Deal. Ε, είμαι και εγώ πολύ φρέσκος. Ε, δεν θα προσπαθήσω να σας δώσω μια συνολική απάντηση. Σας διαβεβαιώ όμως ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο όπως η ψηφιοποίηση και έχουμε όλα τα εργαλεία για να κάνουμε την ε, ανάλυση και τις προβλέψεις που απαιτούνται. Και μάλιστα σήμερα το πρωί ο Χουάννα και εγώ αναφερθήκαμε στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Για τις παραπομπές του ότι δεν σημαίνουν αντίκτυπο, ναι, είναι συζητήσιμο. Εντάξει, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι σημαντικότερα τα έγγραφα πολιτικής και βλέπουμε ότι και σε αυτόν τον τομέα έχουμε αντίκτυπο και βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που εργάζονται στην πράξη χρησιμοποιούν τα έγγραφά μας. Επίσης το ίδιο ερώτημα υπήρξε ακριβώ. Ε, δεν κατάλαβα καλά, για μιλήστε για εξειδίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ, τα πάντα είναι δικής μας σύνταξης, αλλά ε, έχουμε και κάποια έγγραφα εργασίας όπου μπορούν να δημοσιεύσουν ε, με το δικό τους όνομα οι ερευνητές μας. Όσον αφορά την επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, παραδείγματο χάρη θα ξεκινήσουμε στο Ελσίνκι την εβδομάδα κατάρτισης ε, και των σχετικών δεξιοτήτων. Εκπροσωπείται όλη η σχετική κοινότητα, έχουμε κοινά έργα που συζητάμε Όσον αφορά την ε, ποικιλομορφία, αυτό μπορώ να το κρίνω μόνο από την προηγούμενη εμπειρία μου. Είναι η πιο ποικιλομορφή η ομάδα που είχα, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα σπανίως υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα αν είναι καλό ή καλύτερο από ό,τι θα έπρεπε να είναι, δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή. Για τη Βουλγαρία. πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μια λύση για όλους. Ε, πρέπει να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν. Το ΣΕΝΤΕΦΟ προσπαθεί να το κάνει στην ε, προσέγγισή μας με κάθε χώρα που μας πλησιάζει. Και βεβαίως ε, μπορώ να στώσω ένα πρόχειρο παράδειγμα το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει ακριβώς το θέμα αυτό με την μαθητεία και τη σχετική φορολογία. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα, ε, τους ελάχιστους μισθούς ε, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί είναι θέμα των κοινωνικών τέρων. Και Ξέρετε, καμιά φορά είναι τελικά πολύ ακριβές αυτές τι θέσεις και κανείς ε, εργοδότης δεν προσφέρει θέσεις μαθητείας. τέλο. ποια είναι η προσθέμενη αξία μας για τις υπόλοιπε υπηρεσίες ε, και πολλά ακούγονται για την κινητικότητα. Θα πρέπει ε, να γίνεται όπως κάνουν οι φοιτητές με το Εράσμους και εδώ πέρα πάρα πολύ συχνά είναι περιοριστική εθνική κανονισμού. Αυτά τα ολίγα από εμένα. Σας ευχαριστώ και ως κορέλ τελευταίος ευχαριστώ. Εγώ θα κερδίσω το βραβείο για τη συντομότερη παρέμβαση. Η συνεργασία έχει θεμελιώδη σημασία. Και όπως ξέρετε οι διευθυντές ε, των άλλων υπηρεσιών προσκαλούνται ως παρατηρητές στο ΔΣ. Οπότε γι' αυτό το λόγο και μόνο νομίζω πως προχωράει η συνεργασία. Ευχαριστώ. Μπράβο, πραγματικά ε, ήσασταν ο πιο σύντομο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους μας για τις ε, παρουσιάσεις που έκαναν. Πολύ ενδιαφέρουσε, πολλές ερωτήσεις, αλλά ίσως μπορούμε να τα δούμε και κάποια άλλη φορά. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω Καλή σας τύχη και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία. This one was for me, not for you. Okay, so we'll get to the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council amending regulation and... Έχουμε, λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Καλωσορίζω την Κομισιόν, τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Κυρία Σούκοβα, έχετε το λόγο.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 Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να σας παρουσιάσω την πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο εν ώψη δυνατό, πιθανότητας για την άτακτη απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόταση παρά το πρόβλεψη για το Brexit της Κομισιόν και το σχετικό σχέδιο επιφέρει πολύ λίγες τροπολογίες στον κανονισμό. Πρώτα, να σας θυμίσω ότι ο Ευρωπαϊκός, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε το 2007 και αποτελεί έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης για τους εργαζόμενους και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες που έχασαν την εργασία τους λόγω παγκοσμιοποίησης ή λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Με αυτή εδώ την πρόταση η Κομισιόν σηματοδοτεί ότι στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης η ευρωπαϊκή στήριξη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μιας, ενός Brexit άνευ συμφωνίας για τους εργαζόμενους και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες που θα επηρεαστούν από αυτή την απόφαση. Ο στόχος αυτού του ταμείου να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και θα συνεχίσει να παρέχει αυτήν την πολύ χρειαζόμενη στήριξη να, για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν νέε θέσει απασχόληση να ξεκινήσουν νέε εταιρείε. Η τροποποίηση του κανονισ... στον κανονισμό καλύπτει αλλαγή στο πεδίο εφαρμογή τη παρέμβαση, ε, άρθρο 2, ε, παράγραφος 1, ε, όπου ορίζεται το πεδίο της ε, παρέμβασης και εδώ λέγεται ότι η παρέμβαση μέσω του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση μπορεί να ε, ξεκινήσει επί τη βάση της απόσυρσης του, του, Ευρω... Ηνωμένου Βασιλείου από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία ε, εξόδου. Όλοι οι υπόλοιποι κανόνες παραμένουν οι ίδιοι. Δεν, ανα... δεν αυξάνεται ο αριθμός των απολύσεων παραμένουν στους 500 ανθρώπους, δεν αλλάζουμε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του κανονισμού, απλώς ε, επιτρέπουμε στους ανθρώπους που επηρεάζονται από ε, Brexit χωρίς συμφωνία να ε, μπορούν να βοηθηθούν. Επίσης δεν επηρεάζεται ο προπολογισμό, διότι η παρέμβαση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης καλύπτεται από το ετήσιο πλαφόν που είναι 175 εκατομμύρια ετησίως και αυτή η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά και συμμετέχει στην απόφαση για κάθε υπόθεση που, κάθε αίτηση μάλλον βοήθειας από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτά για να ακούσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω την κυρία Σούκοβα, την εκπρόσωπο της Κομισιόν, που, για τις εξηγήσει που μας δίνει σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης λειτουργεί ε, από το 2007, έχει βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους που απολύθηκαν και λειτουργεί πολύ καλά και βεβαίως η κατάσταση ε, αλλάζει και άρα χρειάζεται να προσαρμοστεί και αυτός ο κανονισμός. Ελπίζω ότι θα έχουμε και ένα νέο κανονισμό μέχρι το τέλος ε, του επόμενου έτους. Όπως έχουμε εξηγήσει ε, και έχετε εξηγήσει και εσείς, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προετοιμαστούμε για οποιοδήποτε πιθανή αρνητική επίπτωση που θα δεχτούν οι εταιρείε μας και οι εργαζόμενοι μας λόγω ενός exit δίχως συμφωνία γιατί αυτή η πιθανότητα είναι αληθινή, υπάρχει. Και γι' αυτό και συστήνω να εγκρίνουν τα μέλη της Επιτροπής μας αυτήν σας την πρόταση της Κομισιόν ε, χωρίς άλλες τροπολογίες. Έχω συζητήσει ε, το ζήτημα με όλους τους κοιόδης συζητητές και συμφωνούν μαζί μου. Δεν έχουμε, αρκετό χρόνο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Η έκθεση αυτή πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Οκτωβρίου και την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να εγκριθεί και από την Επιτροπή Απασχόλησης εδώ. Αυτή είναι η κοινή νομοθετική διαδικασία και από γνωρίζω το Συμβούλιο δεν προτίθεται να υποβάλει τροπολογίες σε αυτή την πρόταση. και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, σημαίνει πως και το Συμβούλιο κατανοεί πως πρέπει να τροποποιηθεί αυτός ο κανονισμό μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Άρα τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο οφείλουν να βρουν συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα. Ξέρω ότι ο σκιώδη, η σκιώδης ε, του ΕΛΚ, η κυρία Φλάνση, είχε κάποιες προτάσεις ε, τροπολογίες όσον αφορά αυτό το έγγραφο και θα μας τις παρουσιάσει η ίδια. Αλλά θα ήθελα να σας καλέσω όλους και πάλι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βρούμε μια συμφωνία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε από αυτή την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Νομίζω πως η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μπορεί να είναι αύριο. Να ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση στην Επιτροπή μας στις 2 Οκτωβρίου και ως εισηγήτρια στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν και καλώ όλους σας να τη στηρίξετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη σύντομη εισήγησή σας και τώρα θα δώσω με το λόγο στους κοιόδης. Πρώτα η κυρία Φράνσεν. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που ε, επιμένετε και στο πρόγραμμα. Ε, ήθελα ακριβώ ε, να αναφέρθω στην εφαρμογή του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και ελπίζω πράγματι να μην οδηγηθούμε σε σκληρό Brexit, αλλά αν γίνει αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να είναι έτοιμη 31 Οκτωβρίου να βοηθήσει τα 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους των οποίων οι δουλειές ε, θα κινδυνεύσουν και θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε πάρα πολύ γρήγορα μια απάντηση για να μην είναι και δικό τους ε, το Brexit. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, θεωρούμε να είναι έτοιμο το Ταμείο τον Οκτώβριο και δεν θα υποβάλουμε γι' αυτό το λόγο τροπολογίες στο διατακτικό του κειμένου, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως είπα, για το μέλλον για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοινή δήλωση ζητώντας από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ε, να επιδείξουν την αναγκαία ευελιξία για να βοηθήσουν τους ε, εργαζόμενους για τι βεβαίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οι οποίες είναι η σφονδυλική στήλη της οικονομίας μας πραγματικά κινδυνεύουν από τον Brexit. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί εισηγητρία σας ευχαριστώ για την έκθεση και ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια απάντηση σε όλους τους εργαζόμενους των οποίων η δουλειά ε, κινδυνεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπρόφη από το Ρίνιο και κυρία Φίλιψ. Ετοιμαστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την πρόταση αυτή και την εισηγήτρια. Βεβαίω ε, δεν θέλω να συμβεί το Brexit mm. και θα συνεχίσω να παλεύω να σταματήσει. Το καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα, σε όλα αυτά τα χάλια του Brexit και ενδεχόμενη και τη ζημιά που θα υποστούν οι εργαζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση ατάκτου ε, Brexit. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση είναι χρήσιμο εργαλείο για αλληλεγγύη και για υποστήριξη στους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω παγκοσμιοποίησης ή λόγω οικονομικής ε, κρίσης. Αυτό το ποιοτικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ζωτική σημασία για να υποστηρίξει περισσότερο τους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω των σοβαρών συνεπειών ενός Brexit ατάκτου χωρί συμφωνία. Υποστηρίζω την πρώτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένθερμα και συμφωνώ και με την απόφαση Υγήτρου να μην υποβληθούν τροπολογίε όσον αφορά το νομοθετικό προ... την νομοθετική πρόταση, ούτω ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Υποστηρίζω και τη δήλωση του σκιώδου του ΕΛΚ. Τα κάτι να χρησιμοποιήσουν πλήρω την παρέκκληση που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού στα πλαίσια της, του Brexit, εστιαζόμενοι επί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα πληγούν σκληρότερα Σαν Ευρωβουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, ξέρω ότι το Ταμείο δεν θα είναι διαθέσιμο για εργαζομένου στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, εάν φύγουμε χωρί συμφωνία. Όμω, ελπίζω ότι οσδήποτε πολίτη Ευρω... του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζεται σε άλλο κάτω μέλο, που ίσω χάσει θέση εργασία του λόγω ενό ατάκ του Brexit, θα ωφεληθεί από αυτό το Ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Φίλιπς από τους Πρασίνους και κυρία Λίζη, α ετοιμάζετε, ας προθερμαίνετε. Ευχαριστώ για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πράσινοι ύφο υποστηρίζουν την ταχεία διαδικασία για να εξασφαλίσουμε ότι θα εγκριθεί γρήγορα μέχρι το τέλο Οκτωβριού. Δεν θα υποβάλουμε οποιαδήποτε τροπολογία όσον αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι το κατεπήγον αυτό το ταμείο είναι το κατάλληλο εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί εν τη αυτή περιπτώσει και παρόλο όπως, είπαν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι και εγώ ελπίζω ότι δεν θα λάβει χώρα το Brexit ή τουλάχιστον όχι ε, Brexit χωρίς συμφωνία και η απόστονοτά του δικαστηρίου που ελήφθη τώρα στον Ηνωμένο Βασιλείο που έκρινε ότι ο Πρωθυπουργό μα, ο Μπόρι Τζόνσον, που διέκοψε εργασίε του Κοινοβουλίου, το έκανε αυτό παράνομα. Κατά την άποψή μου, το άτακτο Brexit το κάνει λιγότερο πιθανό. Παρόλα αυτά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Και σωστό είναι αυτό να προχωρήσει το μέτρο όπως προβλέπεται. Υποστεί και στο πεδίο κάλυψης του κανονισμού σε άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει ότι δεν είναι μόνο η παγκοσμιοποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητα αποτελέσματα, όπω η ψηφιοποίηση, η, οικονομία, η μετάβαση οικονομία με χαμηλή κατανάλωση παραγωγή άνθρακα. Πάντα χρειαζόμαστε ένα νέο Green Deal για τη μετάβαση και ένα ταμείο που αμέσω θα υποστηρίζει και που θα χάσουν την εργασία του και θα πληγούν. Το ταμείο δεν έχει σωστό όνομα, αποκαλείται Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και δεν αντικατοπτρίζει πλήρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίο Εργαζόμενο σήμερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λέζε για το ID και η κυρία Σίλουκ ας κάνει προθέρμανση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παραμένει ένα εργαλείο ιδεολογικά επίμαχο. Με αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ανοίξει τα σχήρα τη όσον αφορά τι οικονομικέ και κοινωνικέ καταστροφέ ε, που μπορεί να προκύψουν από την παγκοσμιοποίηση. Η ευθύνη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην έκθεση που παρουσιάζεται σήμερα δεν είναι μικρή και είναι και καρπό αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί την περίπλοκη κατάσταση τη εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σενάριο, το δεχόμενο του Brexit χωρί συμφωνία ε, ε, δημιουργεί αβεβαιότητα και ανησυχίε, Αλλά είναι σίγουρο ότι το Brexit θα έχει βαθιέ συνέπειε κυρίω όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα αρμοδιότητά μα να εξασφαλίζουμε και να υποστηρίξουμε και προωθήσουμε την καριέρα των εργαζομένων που αναπόφευκτα θα πληγούν από ένα Brexit χωρί συμφωνία, αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Ε, η δουλειά του που απειλείται ήδη από την ψηφιοποίηση, από την αυτοματοποίηση και τη ρομποτοποίηση και εν γέννη από την δύναμη τη τεχνολογία. Πρέπει να διαχειριστούμε με τα προσοχή στην ανεργία που προκύπτει την νέα τεχνολογία, επαγρυπνώντα ούτω ώστε η αυτοματοποίηση να είναι πηγή νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και θέσεων εργασία. Υπό το φω αυτών και λαμβάνοντα υπόψη και τα αποτελέσματα τη έρευνα που έχουν δημοσιευτεί που δεν μπορούν να δείξουν τα αποτελέσματα του Ταμείου ήταν θετικά, θεωρούμε θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά αναθεωρήσεων του Ταμείου, μεταξύ αυτών και μια αύξηση του κονδυλίων και μία μείωση του ορίου προσβασιμότητας και έτσι θα είναι ευρύτερο το πλαίσιο κάλυψης των αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής μετάβασης. Τώρα όσον αφορά το επιχείρημα, το θέμα που εξετάζουμε τώρα, δηλαδή η ρήτρα που αναφέρεται ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορέσει να κινητοποιηθεί σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, με κριτήρια που προβλέπονται και πρέπει να γίνονται σεβαστά. Πρέπει να γίνει αυτό και τα, εάν βγει το, το Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγηθεί σε αλλαγή η αγορά εργασία και η ενιαία αγορά και θα έχει αντίκτυπο διαφορετικό σε κάποιου οικονομικού τομεί και κάποιε περιοχέ. Και η ΛΕΓΑ και η ID θα φροντίσει στην Ιταλία να μην χαλεί ούτε μια θέση απασχόληση στα πλαίσια του Brexit χωρί συμφωνία και θα πρέπει να υπάρξει συνεχής έλεγχος ε, της ε, κατάστασης ώστε να υπάρχουν ενεργά μέτρα όσον αφορά την αγοργασία που σκόπο θα έχουν την επανένταξη σε ποιοτική απασχόληση στους τομείς και στις περιοχές της Ιταλίας θα πληγούν περισσότερο. Κλείνοντα, η αντιπροσωπεία μα υποστήριξε και υποστηρίζει τι παρεμβάσει του εργαλείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θεωρεί ότι είναι μερική αποζημίωση για τους συμπολίτε και τους εργαζομένους μας. Γι' αυτό το λόγο θα εξολογήσουμε και τις τροπολογίες που προβλέπουν τη θέσπιση μιας ρήτας που, που λέει ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορεί να κινητοποιείται και σε περίπτωση Brexit No Deal. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για το χρόνο που μου δώσατε. Λάβαμε ένα μήνυμα από τους διερμηνείς, αν μπορείτε να μιλάτε πιο αργά, πιο αργό ρυθμό, παρόλο που ξέρω που εγώ σας πρόχνω, σας πιέζω χρονικά. Για το ECR, η κυρία Σίντλο και ο κύριος Γκουσμάου μετά. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο για την Προσωπική στην Παγκοσμιοποίηση δεν δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους εργαζομένους που πλήττονται από περιστάσεις ανεξέλεγκτες από αυτούς. Το Brexit σίγουρα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Διότι δεν θα πλήξει μόνο τους εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ευρωβουλευτής, αλλά όπως ίσως κάποιοι από εσά γνωρίζουν, είμαι πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας. Και Είχα πολλές δυνατότητες να συνομιλήσω με τους συμπολίτες μου. Πολλοί από αυτούς ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκείνοι οι Πολωνοί που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο επί τρία χρόνια ανησυχούν και πιέζονται γιατί δεν ξέρουν πώς θα επηρεάσει το Brexit τη ζωή τους και την εργασία τους. Δεν ξέρουμε τι Brexit θα αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό ως σκιώδης για το ECR όχι μόνο υποστηρίζω αυτή την πρόταση, αλλά θα ήθελα να κάνω και άλλη μια πρόταση. Προτείνω να επεκτείνουμε το κείμενο και να πούμε ότι το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν η έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση έχει αρνητικέ συνέπειε. Δηλαδή, να μην λέμε ότι μόνο σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρί συμφωνία, αλλά να αντιμετωπιστούν οι αρνητικέ συνέπειε του Brexit εν γέννη. Έτσι, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ανταποκριθούν κατάλληλα σε ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν. Κυρίε και κύριοι, αυτό το ταμείο ήδη έχει βοηθήσει 150.000 πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω ότι το Brexit είναι ακόμα μια δυνατότητα, δεν μπορούμε να διαγράψουμε αρνητικές συνέπειες αυτού, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες από τις αρνητικές συνέπειες και να προετοιμαστούμε για παν ενδεχόμενων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκουε, κύριε Γκουσμάου. Αλλά πού είναι ο κύριος Γκουσμάου, δεν τον βλέπω. Α, δεν είναι εδώ κάποια μέλη, ο κ. Πάτρος Λέναρτς και η κυρία Αντριένε θέλουν να λάβουν το λόγο. Ο κ. Μπάτν πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζει να μ' αρέσει το και να το συνηθίζω το Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και θα δαπανίσει 50% περισσότερα ιδιωτικά ε, τζετ για τους γραφειοκράτες Πρέπει να κάνουμε περισσότερο για το Ιράν, αλλά δεν διευκολύνει την αντιπροσωπεία τη στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν υπεύθυνη για Brexit χωρί συμφωνία, αλλά το ψήφισμα πολλοί από εσά ψηφίσατε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο επιμένει επί του Ιρλανδικού backstop και κάνει το no deal σχεδόν από αυτό Και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει περισσότερα χρήματα των μελών, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, για να υπάρξει αποπληρωμή δεν υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό ε, ακούει πολλέ επικρίσει του Ταμείου Προσαρμογή και Είναι άδικο και αθέμητο στοχεύει σε μεγαλύτερους οργανισμούς, αλλά είναι άπελπης προσπάθεια για μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και μικροεπιχειρηματίες που είναι 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είναι άκρο αναποτελεσματικό, είναι αδύνατο να αξιολογηθεί κατά πόσο οι εργαζόμενοι που λάβανε βοήθεια από αυτό το ταμείο είναι καλύτερα όσον αφορά την προσπάθειά του να βρουν δουλειά από εκείνου που δεν πήραν καθόλου χρήματα. Πολλά κράτη-μέλη επανειλημμένα καταψήφισαν αυτό το ταμείο, ισχυριζόμενο ότι δεν δίνει αξία για τα λεφτά του και δεν δεν αξίζει τι επενδύσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνει τη διαφορά σχέση με το εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι αρχικά δημιουργήθηκε το Ταμείο για να παράσχει υποστήριξη στην παγκοσμιοποίηση ε, για μεγάλε οικονομικέ αλλαγέ, αλλά δεν νομίζω ότι δημιουργήθηκε ε, όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα από δράσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και δεν πιστεύω καν λεπτό ότι το Brexit μπορεί να συγκριθεί με γεγονότα όπως είναι το οικονομική, οικονομική του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τα χρήματα των ε, κρατών μελών για να υποστηρίξει και να αποσβέσει τα αρνητικά αποτελέσματα κρίσεων που ήδη δημιουργεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέναρς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Brexit είναι ούτως ή άλλως μια κακή ιδέα και βεβαίως μόνο οι τιμένους θα έχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά ένα Brexit χωρίς συμφωνία είναι ε, η μητέρα όλων των κακών ιδεών και θα προξενήσει ζημίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, βέβαια ο προηγούμενος ομιλητής ε, έκανε την σύγκριση με την οικονομική κρίση που κόσσε 500.000 θέσει εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από ένα εκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α τα πει αυτά, α τα εξηγήσει στους ε, ψηφοφόρους τους. Δηλαδή το να λέμε ότι ας γίνει ό,τι θέλει και 1,2 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι εκ των οποίων 300.000 ε, στην Ολλανδία, την χώρα μου γιατί, γιατί φοβούνται και σκέφτονται βράχη πρόθεσμα οι λαϊκιστές και οι μπρεξτρεμιστές. Λοιπόν, θα πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βετρένεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εισηγήτρια για την εργασία της, αλλά και το σύνολο των σκιωδών εισηγητών. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, όταν λέμε ότι αυτή η πρόταση είναι θεμελιώδης και πρέπει να την υιοθετήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Το κείμενο αυτό είναι απόδειξη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για όλες τις καταστάσεις και προβλέπει τις συνέπειες του Brexit. Χάρη σε αυτή την τροπολογία, τροποποίηση μάλλον, ε, θα μπορούμε από το 2020 να βοηθήσουμε ε, τους εργαζόμενους που είναι θύματα αναδιάρθρωσης ε, εταιριών, εάν υπάρξει τελικά το, γίνει το Brexit και αν γίνει μάλιστα Brexit χωρίς συμφωνία. Αυτό ε, σημαίνει ότι θα, υπάρχει σημαντική, ε, θα, σημαντικός στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, δείξουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση. Στη Γαλλία και στην περιφέρειά μου τη Βρετάνη, πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι ε, θα υποστούν αυτές τις συνέπειες, γι' αυτό είναι επίγον και ευχαριστώ τους συναδέλφους που το έκαναν να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση όσο γίνεται πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια ώστε να μπορέσει και εκείνη να αντιδράσει σε συζήτηση και στην ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές που υπέβαλαν τις απόψεις τους ε, ε, ε, γνώμες ε, πρέπει να στηρίξουμε όντως την πρόταση της Επιτροπής γιατί όπως είπα είναι μια θέση που στηρίζεται και από το Συμβούλιο για να έχουμε μια γρήγορη λύση Ο κανονισμός είναι υπό αναθεώρηση θα έχουμε νέο κανονισμό του χρόνου και θα έχουμε και καλύτερες δυνατότητες για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους μας. Ευχαριστώ και εγώ ε, μια σύντομη αντίδραση από πλευρά της Κομισιόν. Μάλιστα, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που στηρίζουν την ε, πρόταση της Κομισιόν. Ε, προσβλέπω στο να συζητήσουμε τον